Καλησπέρα σας. Προτείνω να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε γεμάτη μερίσια διάταξη. Καθώς είναι η τελευταία μας εβδομάδα. Καλωσορίσατε λοιπόν όλοι. πριν ζητήσουμε από τη Βελγική Προεδρία να μας ενημερώσει για τις προτεραιότητες της, προτείνω να προσθέσουμε ένα σημείο στην ημερήσια διάταξη τη σημερινή. Το ζήτησαν οι φιλελεύθεροι, οι γκούε, οι S&D και οι πράσινοι. Αφορά τους μετανάστες στην Λιβύη. Το αναφέραμε και στο Στρασβούργο. Όσον αφορά τη Μολδαβία, θα συζητήσουμε το θέμα μετά την παρέμβαση του Επιτρόπου. Ελπίζουμε ότι αύριο στην παρέμβαση του Επίτροπος Δεγκούχτ θα μας δώσει την απάντηση. Άλλη μία ανακοίνωση και περνάμε στην, στο κύριο μέρος της συνεδρίασης. Μετά από πρόταση των συντονιστών προτείνω να δεχτούμε τους εξής ε, εισηγητές. Την Άννα Γκόμες, που δεν την βλέπω εδώ, για την ανακοίνηση για τα CBR, ε, τα, το σχέδιο δράσης δηλαδή για τις ουσίες CBR και τον ε, κύριο Κίρχοπ για την ε, συμμετοχή Ελβετίας, ε, Ισλανδίας, Νορβηγίας και Λίχτενστάιν για την ανάπτυξη του κεκτημένου Σέγγεν. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρούμε ότι γίνονται δεκτά όλα αυτά και μπορούμε να περάσουμε το βασικό περιεχόμενο της συνεδρίασης, σημείο 3. όχι. Όχι, δεν έχω πρόβλημα με τις ανακοινώσεις σας μέχρι τώρα, αλλά πριν ε, περάσουμε στο σημείο 3 θα ήθελα να αναφέρω κάτι ακόμη για την ημερήσια διάταξη. Για την αυριανή ημερήσια διάταξη. Για την υπόθεση Βίσκε και Ερυθρέας έχουμε ζητήσει και από την Μάλστρομ και από τη τον Φιουλερ μία απάντηση. Δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση από τον Φιουλερ και επειδή αυτό το θέμα αφορά και την πολιτική γειτονία και την μεταναστευτική πολιτική, θα ήθελα να ζητήσουμε να έλθει και ο κύριος Φούλερ αύριο εδώ. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Ε, κυρία Πρόεδρε, δεν έχουμε καμία ενημέρωση επί του θέματος. Άρα Όποτε θέλουμε να προσκαλούμε επιτρόπους σε μία συνεδρίαση θα πρέπει τουλάχιστον να έχουμε κάποια ενημέρωση για το τι θα συζητηθεί. Δεν μπορούμε να λέμε θα μιλήσουμε για πολίτες της Ερυθρέας στη Λιβύη ή για Σομαλούς στην Ελλάδα και αυτό είναι όλο. Πρέπει να γνωρίζουμε και ποιο είναι το περιεχόμενο αυτή της συζήτησης να γνωρίζουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται και έτσι να αποφασίζουμε για το αν θέλουμε να προσκαλέσουμε τον Επίτροπο συνεδρίαση ή όχι. Καταρχάς, όπως είπα, υπήρξε αίτημα από αυτές τις πολιτικές ομάδες που ανέφερα. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, να πω ότι ναι, δέχομαι τις επικρίσεις σας, αλλά ζήτησαν αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη φιλελεύθερη πράσινη κούε και σοσιαλιστές. Για το δεύτερο σημείο, για τον κύριο Φίλερ, ήρθαμε σε επαφή με τη γραμματεία του και μας είπαν ότι θα επανέλθει στις 14 δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς θα απαντήσει, όμως γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ασχολείται με το πώς θα αντιμετωπίσει το θέμα. Πάντως η ΛΥΜΠΕ δεν θα μπορέσει να έχει συνεδρίαση για αυτό το θέμα τότε. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε και ελπίζουμε να έχουμε περισσότερες ε, πληροφορίες στη συνέχεια. Θα δώσω τώρα το λόγο στον ε, Υπουργό, τον κύριο Ντεκλέρκ, να μας ενημερώσει για τις προτεραιότητες της Βελικής Προεδρίας στον τομέα της δικαιοσύνης. Με την ε, συνθήκη της Λισαβόνας προφανώς υπάρχουν πολλά νέα στον τομέα αυτό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Θα μιλήσω Ολλανδικά, που είναι και η μητρική μου γλώσσα. Ευχαριστώ. Είναι για μένα μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα ενώπιόν σας. Και ακριβώς αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή έχει ιδιαίτερη δυναμική και έχει μεγάλο έργο επιτελέσει. Και είχα ήδη την τιμή σε σχέση με την συμφωνία που είχε επιτευχθεί να έχω επαφές με τα μέλη της Επιτροπής σας και την προηγούμενη εβδομάδα είχα επίσης την τιμή να παρίσταμε στις συζητήσεις στην Ολομέλεια στην περίοδο συνόδου του Ιουλίου στο Στρασβούργο ευχαριστώ επίσης θερμά την Πρόεδρο για το ότι συνεργαστήκατε να επιτευχθεί μια συμφωνία και ευχαριστώ επίσης και τον εισηγητή κύριο Άλβαρο. Είναι πραγματικά μια εξαιρετική έκθεση και είναι πραγματικά καλό το ότι είχατε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους εμπλεκόμενους. Ναι, κατά τη διάρκεια φυσικά της Βελγικής Προεδρίας θα πρέπει να προβληματιστούμε για το κατά πόσον το πρόγραμμα της Στοκχόλμης μπορεί να αποκτήσει σάρκα και οστά και να αναζωογονηθεί. Υπάρχουν φυσικά προτεραιότητες που έχουμε και κάποια στοιχεία μπορώ να σας αναφέρω. Δεδομένου επίσης και το ότι μια συζήτηση θα ήθελα να διεξαχθεί ώστε να επιτευχθεί πρόοδος επί των θεμάτων αυτών. Φυσικά συνεχίζουμε, είναι αυτονόητο αυτό, στα όσα επετέλεσε η Ισπανική Προεδρία με τη δική της ξεχωριστή δυναμική και είναι εδώ εντολή να υπάρξει συνέχεια και συνέπεια και συνεκτικότητα. Δεν πρόκειται μόνο για α, κάποια θέματα αλλά για συνέχεια και συνεκτικότητα και ελπίζω ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε. Τρία στοιχεία θα ήθελα να αναφέρω τα οποία θα θέλαμε να υλοποιήσουμε. Το πρώτο σημείο ποιο είναι. Είναι για μας φυσικά παραδοσιακά πολύ σημαντικό και είναι η θεματολογία που αφορά την προστασία των θυμάτων προστασία των θυμάτων εγκλημάτων. Και στο παρελθόν στο Βέλγιο ήταν μείζον θέμα για μας και το τονίζαμε πάντα. Θέλουμε λοιπόν πραγματικά τα θύματα να βοηθηθούν. Εκείνοι οι οποίοι είναι οι πιο ευάλωτοι, τα παιδιά για παράδειγμα, και τα οποία <clears throat> την χάνουν κακομεταχείρισης και κακοποίησης με την παιδική πορνογραφία. Είναι ένα θέμα το οποίο σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να αντιμετωπιστεί και σε σχέση με ε, ορισμούς και θέματα είναι κάτι διασυνοριακό φυσικά. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι ευχαριστούμε καταρχήν θερμά την Ισπανική Προεδρία και θέλουμε να συγχαρούμε την Ισπανική Προεδρία για τις δραστηριότητες της, για τις ε, προσπάθειες ε, να υπάρξει ένα πλαίσιο για την προστασία αυτών των ατόμων. Τους τελευταίους μήνες υπήρξε πρόοδος για τα μέτρα προστασίας που στα διάφορα κράτη-μέλη θα υλοποιούνται. Η Βελγική Προεδρία θέλει να εμβαθύνει περισσότερο σε αυτό και θα είναι και μια προτεραιότητα και από πλευρά μας και δική σας. Θέλω να ευχαριστήσω και σε σχέση με την Προεδρία που δίνεται η δυνατότητα να εμβαθύνουμε σε σχέση με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, την ΛΥΜΠΕ, και για την οδηγία για την προστασία, όπως είπα, των θυμάτων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το μέσο εδώ να χρησιμοποιηθεί και να πάρει συγκεκριμένα σάρκα και οστά. Και αυτό όχι μόνο σε σχέση με τους συναδέλφους του Συμβουλίου που πρέπει να πιστούν ώστε να υπάρξει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δράσης, αλλά θα προσπαθήσω και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταλήξουμε σε συμφωνίες, σε, μια πρώτη, σε πρώτη ανάγνωση για αυτό το, προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα με το εμπόριο ανθρώπων φυσικά, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες να υπάρξει μια κοινή κοινοτική πολιτική στην οποία θα καταλήξουμε για να καταπολεμήσουμε την εκμετάλλευση την σεξουαλική και την κακοποίηση των παιδιών και την να καταπολεμήσουμε και την παιδική πορνογραφία και θέλουμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής σας Επιτροπής στο δυνατόν πιο νωρίς. Και ένα άλλο κέντρο βάρους που θα θέλαμε να θέσουμε. Είναι η δικαστική συνεργασία, η συνεργασία όσον αφορά τα δικαστικά θέματα. Να βελτιωθεί αυτή η συνιστόσα. Και με την καταπολέμηση του εγκλήματος. Περισσότερο από οποτεδήποτε πρέπει εδώ πραγματικά να συνεργαστούμε. Η συνεργασία όσον αφορά τα δικαστικά θέματα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ενδυναμωθεί, ώστε να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα πρέπει πραγματικά να καταβάλουμε προσπάθειες να υλοποιηθούν οι στόχοι. Και είναι πρόδειλο, είναι προφανές ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε και τους, ε, τις αποφάσεις ε, και ε, της, ε, την μέρημνα που λαμβάνουν οι δικαστές. Πρέπει να πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Για τη Βελγική Προεδρία είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα από τη διαδικασία της αμοιβαίας αναγνώρισης να προχωρήσουμε. Και πρέπει μεθοδολογικά να εκπονήσουμε τις αρχές εκείνες που θα ακολουθούνται. Απλούστευση, ενιαιο, ενιαιοποίηση, ένα ενιαίο, ενιαίο πιο ενιαίο, ε, ομοιογενές πλαίσιο. Και φυσικά όλα αυτά πρέπει να υλοποιούνται και να εκτελούνται. Και εδώ είναι σημαντικό να δούμε ποιες χώρες, ποια κράτη συγκεκριμένες εξελίξεις ε, ε, ακολουθούν αυτές τις εξελίξεις και κινητοποιούνται. Πρέπει και από πλευρά του Συμβουλίου να εγγραφεί το θέμα στην ημερήσια διάταξη και στην ημερήσια διάταξη των Υπουργών Δικαιοσύνη. Και η αμοιβαία νομική αρρωγή, η συνδρομή, είναι και αυτό ένα πεδίο συνεργασία όπου χρειαζόμαστε τη συνεργασία αυτή και από κοινού με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Υπάρχει μια ομάδα κρατών μελών και το Βέλγιο εδώ έχει αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να καταλήξουμε σε μια ευρωπαϊκή εντολή έρευνας ή ένα ένταλμα ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όσον αφορά τεκμήρια και πιστήρια που θα αναγνωρίζονται αμοιβαία σε σχέση με τα δικαστικά θέματα. Αυτό το μέσο είναι πολύ σημαντικό, ώστε πολύ γοργά να υπάρξει τυποποίηση, να υπάρξει προώθηση των ανακριτικών δράσεων και των ε, ερευνών ώστε να μπορούμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα μέσω ανακριτών ή μέσω ερευνητικών δράσεων δικαστικών αρχών. Με αυτό το μέσο θα μπορέσουμε να δώσουμε απάντηση σε συγκεκριμένες ανάγκες και φυσικά τα δικαιώματα των εμπλεκόμενων να μπορούν να αντιμετωπιστούν σωστά. Εδώ η Βελγική Προεδρία θέλει να δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα, να προχωρήσει αυτή η πρωτοβουλία και από κοινού με τα κράτη-μέλη να ευδοκιμήσει. Ένα περαιτέρω σημείο το οποίο σύντομα θα ήθελα να αναφέρω σε σχέση με αυτά, μια και το Σεπτέμβριο θα διοργανώσουμε ένα σεμινάριο στην πόλη Μπρούγκε, είναι το ότι πρέπει να διαπιστώσουμε ότι πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό ε, εμπλεκόμενο στο δικαστικό επίπεδο στην ευρωπαϊκή, στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για την ε, συνδρομή και το πλαίσιο το οποίο θα θέλαμε να θεσπιστεί ώστε να εξεταστούν τα θέματα ανακριτικών ε, πρωτοβουλειών και το θέμα της Eurojust είναι σημαντικό και για τους ε, εισαγγελείς ε, και για το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο. Νομίζω ότι πραγματικά φιλόδοξα πρέπει να προχωρήσουμε με φιλόδοξους στόχους. Είμαι πισμένος προσωπικά ότι κατά τούτο θα έχουμε μια καλύτερη δυνατότητα παρακολούθησης των ποινικών αυτών θεμάτων και δίωξη των ε, εγκληματιών. Θέλουμε να υπάρξει η δυνατότητα να δούμε πώς δίνουν, δίνονται δυνατότητες, διανοίγονται δυνατότητες από τη συνθήκη της Λισαβόνας όσον αφορά τις ε, δράσεις ε, εισαγγελιών και εισαγγελέων. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διερευνήσουμε ώστε με τους Υπουργούς Δικαιοσύνης ε, να καταλήξουμε και να προβληματιστούμε σε συγκεκριμένη θεματολογία. Αποκινούμε την δικαστική συνεργασία. Είμαι πεισμένος ότι στην καθημερινή ζωή χρειαζόμαστε αυτή τη συνεργασία. Ιδιαίτερα σε συνοριακές μεθοριακές περιοχές. Οι άνθρωποι που ζουν στις μεθοριακές περιοχές γνωρίζουν ότι είναι σημαντικό διασυνοριακά να δρούμε και να δράσουμε και ευρωπαϊκά, πανευρωπαϊκά, ενωσιακά να κινητοποιηθούμε πρέπει στην πρακτική εφαρμογή καθημερινά όλα αυτά να είναι λειτουργικά και να μπορούν ε, να εφαρμοστούν. Και η Βελγική Προεδρία θα ήθελε να διοργανώσει ένα σεμινάριο ώστε να προαχθούν αυτοί οι στόχοι. Μια άλλη προτεραιότητα τώρα είναι η προσπελασιμότητα των ε, δικαστικών θεμάτων και των θεμάτων δικαιοσύνη. Θέλουμε να έχουμε περισσότερε εγγύσει, περισσότερα χέγγια για του πολίτε. Η προσχώρηση τη Ευρωπαϊκής Ένωσης στην, Ευρωπαϊκή, στην Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είναι μια ενδυνάμωση για τα δικαιώματα των πολιτών. Και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια θετική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο τη Ευρώπη, Όσον αφορά και τα δικαιώματα των όσων εμπλέκονται σε ποινική δικαστικές ε, ε, διαδικασίες και σε δίκες θέλουμε να υπάρξουν ελάχιστες προδιαγραφές που θα ε, θεσπιστούν όσον αφορά μεταφραστικό έργο και διερμηνία. Είναι πολύ σημαντική αυτή η σύνδρομη όσον αφορά τους εμπλεκόμενους σε ποινικέ διεργασίες και για τους υπό ανάκριση ευρισκόμενους. Εδώ αναμένουμε πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζουμε ότι θα σημειωθεί πρόοδος. Τα κράτη-μέλη έχουν εδώ εκφράσει τα ε, ε, ε, αιτήματά τους, τα μελήματά τους και αυτό είναι σημαντικό. Όσον αφορά τις πτυχές του αστικού δικαίου πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια ώστε οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ακολουθηθούν που θα βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των πολιτών και που και στην νομική επιτροπή, στην Γιούρη, θα υπάρξει ενημέρωση. Θα ήθελα όμως εδώ να υπάρξει πρόθεση αυτών των θεμάτων είναι πολύ σημαντικό διότι όταν υπάρχει ευρωπαϊκή προστασία όταν όλα τα μέτρα ε, μέσα συνδρομής ε, θέλουμε να υλοποιηθεί χρειαζόμαστε την e-justice, ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Είναι μια περαιτέρω συνεισφορά για την προσπελασιμότητα στα θέματα δικαιοσύνης για όλους. Και η δυνατότητα βίντεο διασκέψεων ή ηλεκτρονικών υπογραφών και κωδικών ή ε, την δυνατότητα μητρώων ή μητρώων σε σχέση με αφαιρεγγιότητα. Ελπίζω ότι αυτή την εβδομάδα μέχρι τις 16 ε, Ιουλίου θα υπάρξει ε, πρόθεση και από από το άτυπο συμβούλιο να υπάρξει ένα ε, ένας πυλώνας ε, πορτάλ ε, για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη e-justice. Εδώ και οι συναφείς προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και οι πρόεδροι της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και Πολιτικών Ελευθεριών λένε και Λόπεθ Αγγιλάρ θα μπορέσουν να εμπλακούν. Θέλουμε να υπάρχει προσπελασιμότητα για όλους τους πολίτες της Ευρώπης να μπορεί να υπάρξει συμμετοχή και εμπλοκή όσον αφορά τα νομικά μέσα και τις δυνατότητες ώστε να μπορούν οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις νομικές δυνατότητες. Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια να εφαρμοστούν αυτά και να αποκτήσουν ε, σάρκα και οστά και να είναι διαθέσιμα στους πολίτες. τώρα όσον αφορά τις διατλαντικές σχέσεις. Για αυτές τις διατλαντικές σχέσεις μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να πούμε ότι είναι σημαντικό στο Συμβούλιο έχουμε και την εντολή διαπραγματεύσεων που εγκρίναμε όσον αφορά μια γενική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΕΠΑ ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Μέσα στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντική και η συμφωνία SWIFT για την διάθεση στοιχείων στις ΕΠΑ. ΕΕ. Είναι εδώ ένα φιλόδοξο μέσο ε, το οποίο ε, δημιουργείται για την ε, δράση σε αυτό το πεδίο. Και είναι ενδιαφέρον να δει κανεί ε, και την ε, αντίδραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εν κατακλείδη συνοψίζοντα θα ήθελα να πω το εξή. Φυσικά έχουμε μεγάλε φιλοδοξίε Πιστεύουμε όμως από την άλλη πλευρά ότι πρέπει να διασφαλίσουμε τη συνέχεια και συνεκτικότητα. Να υπάρχει καλή επικοινωνία με την Επιτροπή αυτή και είμαστε πισμένοι ότι μπορεί να σημειωθεί πρόοδος. Σας διασφαλίζω ότι τα μηνύματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν γίνει αντιληπτά, έχουν, γίνει, έχουν κατανοηθεί όσον αφορά και τη μεθοδολογία και τις συμφωνίες μαζί σας με το Συμβούλιο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτή νομίζω είναι η σωστότερη μέθοδος ώστε να σημειώσουμε πρόοδο πρόοδο, πρόοδους όσον αφορά την Ευρώπη και τα, ε, δικαιοσύνης και την προστασία των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω ερώτηση. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Φαίνεται ιδιαίτερα φιλόδοξο το σχέδιο σας και υποθέτω ότι θα έχουμε και πολλούς ερωτήσεις από τους συντονιστές και τα υπόλοιπα μέλη. Ξεκινάμε με τον κύριο Μπουσουτήλη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον Υπουργό που ήρθε σήμερα στην Επιτροπή μας και σας ευχαριστούμε για τις ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες που αναφέρατε όσον αφορά το έργο της Προεδρίας σας. Μία ερώτηση. Είπατε ότι η Προεδρία σας ενδιαφέρεται να ασχοληθεί και να προχωρήσει με το ευρωπαϊκό ένταλμα αποδείξεων, evidence order. Γνωρίζετε κύριε Επίτροπε ότι του τελευταίους μήνες είχαμε κάποια προβλήματα και διαφωνίες μεταξύ Επιτροπής και Συμβουλίου όσον αφορά τέτοιου είδους συμφωνίες που είχαν εγκρίνει κάποια κράτη-μέλη. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν η Προεδρία έχει συζητήσει το θέμα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με την πρότασή σας. Αν σκοπεύετε να προτείνετε μια κοινή θέση με την Επιτροπή, αν περί αυτού πρόκειται γιατί γενικά θα ήθελα να βλέπω περισσότερη αρμονία μεταξύ Κομισιόν και Συμβουλίου. Ε, εσείς δεν θεωρείτε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό το θέμα όπως ακριβώς ε, και το ευρωπαϊκό ένταλμα. Θέλουμε λοιπόν να συνεργαστούμε μαζί σας και να συνεργαστούμε πλήρως και με την Επιτροπή για να καταλήξουμε σε μία πρόταση που θα είναι και στους δύο ευπρόσδεκτη. Τα σχόλια σας επ' αυτού λοιπόν θα ήθελα να ακούσω. Ευχαριστώ. Προτείνω να ακούσουμε δύο-τρεις ερωτήσεις από μιλητές και μετά να δώσουμε το λόγο στον Υπουργό. Η Κάρμελ Λόπες, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών. Κάρμεν, θες να κάνεις ερωτήσεις εκ μέρους των Σοσιαλιστών. Ναι, παρακαλώ. Sí, gracias, señora presidenta. Sí. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εμείς ε, ενδιαφερόμαστε να μάθουμε μερικές ε, λεπτομέρειες παραπάνω γύρω από ζητήματα τα οποία παρέμειναν εκκρεμή μετά την Σουηδική και την Ισπανική Προεδρία. Πρόκειται για την σώματεμπορία γυναικών και το πρόβλημα των ανηλίκων. Και θα ήθελα επίσης, επειδή και ο συνάδελφος Μπουσούτιλ επέμεινε σε αυτό, να μας πληροφορήσετε σχετικά με το θέμα της βίας κατά, το, κατά των γυναικών δεν έχουμε στατιστικές, δεν έχουμε στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά. Θα θέλαμε λοιπόν οι ευρωπαϊκές χώρες να προχωρήσουν περισσότερο στη μελέτη αυτού του προβλήματος αλλά και στον ορισμό αυτής της βίας κατά των γυναικών. Δεν υπάρχει οδηγία για αυτό το θέμα. Οπότε οι ευρωπαϊκές δυνάμεις ασφαλείας εργάζονται με μηχανισμούς κατεπήγοντος για αυτό το θέμα. Ρωτώ λοιπόν, θεωρεί η Βελγική Προεδρία ότι κατά την Προεδρία της θα εξετάσει αυτό το ζήτημα με όλες τις ε, ε, επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν και θα το προχωρήσει το θέμα αυτό. Θα ζητήσω από τον Υπουργό να απαντήσει στις δύο ερωτήσεις αυτές καθώς σχετίζονται μεταξύ τους. Ευρωπαϊκό ένταλμα προστασίας και διαφωνία Επιτροπής και Συμβουλίου. Πώς αντιμετωπίζετε αυτά τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ. Είναι μια ουσιοδέστατη ερώτηση σε σχέση με την συνέχεια που πρέπει να διασφαλίσετε. Το πρώτο σημείο αναφερόταν σε αυτό το ένταλμα ανακρίσεων αλλά και το ένταλμα των τεκμηρίων ή αποδείξεων είναι συζήτηση που συνεχίζεται και θα συνεχιστεί. Θέλουμε όμως και μια ευρωπαϊκή ανακριτική εντολή. Εδώ πρέπει σε ένα σφαιρικότερο πλαίσιο να ενταχθούν αυτά τα θέματα και θέλουμε και ένα τυποποιημένο πρότυπο να ακολουθηθεί. Το τονίζω, είναι μια πρωτοβουλία που ε, έχει αναλυφθεί και μια σειρά χωρών έχουν αρχίσει ήδη να προωθούν αυτά τα θέματα. Με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε ήδη συζητήσει εκτενώς και διεξοδικά το θέμα και επιβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η επικοδομητική θέση υιοθετείται εναντί αυτών των πρωτοβουλειών. Και τώρα αυτό το οποίο λέμε είναι ότι αυτά με αρμονικό τρόπο θα προχωρήσουν με ένα εναρμονισμένο τρόπο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, αλλά φυσικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εμπλακεί και να συνοδεύσει αυτά τα θέματα. Πρέπει με κοινέ σκέψεις και προβληματισμό να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε δράση. Ε, και για το SWIFT, όπως είχε, υπήρξαν οι τοποθετήσεις, πρέπει να δούμε ποιες πρωτοβουλίες μπορούν να αναλυθούν σε, αυτή σε αυτόν τον τριπλό άξονα για την εντολή, για παράδειγμα για τα τεκμήρια, evidence order, χρειάζονται διαβουλεύσεις πώς αυτά μπορούν να υλοποιηθούν από κοινού με το investigation order, με την ερευνητική ή ανακριτική δράση. Εδώ υπάρχουν επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε πώς από τεχνικό επίπεδο σε πολιτικό επίπεδο μπορούν αυτά να οριμάσουν και να προαχθούν. Αυτά τα οποία αναφέρθηκαν από την ε, συνάδελφό σας ε, κυρία Λόπεθα ε, αφορούν μια σύνθετη προβληματική παράδειγμα το εμπόριο ανθρώπων αλλά παράδειγμα και τα παιδιά τα προβλήματα που αφορούν τα παιδιά Ιδιαίτερα τονίζονται αυτές οι πτυχές και υπάρχουν και αντίστοιχες νέες πρωτοβουλίες και θέλουμε με προτεραιότητα να αντιμετωπιστούν αυτές οι πρωτοβουλίες. Να υπάρξει μια κοινοτική προσέγγιση, ενωσιακή προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη δική σας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Αυτό θέλουμε να επιτύχουμε και από κοινού με την Προεδρία μας μπορούμε και με εσάς να συνεργαστούμε για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Το θέμα του εμπορίου ανθρώπων θα πρέπει και αυτό να αντιμετωπιστεί η κακοποίηση ε, των παιδιών ήδη στην εισαγωγή μου επεσήμανα αυτή την προβληματική, αυτή τη θεματολογία, την κακοποίηση των παιδιών και τα θέματα του διαδικτύου και υπάρχουν νέες πρωτοβουλίες που έχουν προαχθεί, που έχουν προωθηθεί θέλουμε αυτά, αυτές οι πτυχές να μεγιστοποιηθούν ε, να βελτιστοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν. Αλλά πρέπει και τη συνέχεια και συνεκτικότητα να λάβουμε υπόψη. Δεν είναι τίποτα καινούριο. Εμεί ω ε, Βελγική Προεδρία υποστηρίζουμε αυτέ τι πρωτοβουλίε που είχαν αναλυφθεί και είμαστε πεισμένοι ότι είναι σημαντικέ ε, πρωτοβουλίε. Μια άλλη πτυχή είναι τα θέματα προστασία. Και εδώ με την Ισπανική Προεδρία υπήρξε και από πλευρά μα πάντα υποστήριξη αυτή τη με ένα νέο ανανεωμένο τρόπο πρέπει να μπορέσουμε να, να το εξετάσουμε με λεπτομέρειες, με νομικές ε, ας το πτυχές που θα ε, φωτίζουν κάποια θέματα για τα, τις εγκληματικές ε, πτυχές που αφορούν το θέμα το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνη θα εγγράψει αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη των εργασιών του. Όταν θα συνέλθει, αυτό το θέμα θα τύχει ιδιαίτερη προσοχή και ελπίζουμε ότι θα έχουμε μέγιστη υποστήριξη των κρατών μελών μέγιστη υποστήριξη για ένα προσαρμοσμένο κείμενο το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις τεχνικές πτυχές και μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να ενισχύσουμε, να ενδυναμώσουμε την συνέχεια και συνεκτικότητα και να διασφαλίσουμε την πρόοδο, ιδιαίτερα όσον αφορά και την ε, το ένταλμα προστασίας. Είναι κάτι σημαντικό που έγινε από την Ισπανική Προεδρία και ε, επίσημα και τυπικά τον Οκτώβριο θα πρέπει στο μέτρο του δυνατού, στο μέτρο του εφικτού να ολοκληρωθούν αυτές οι δράσεις για να καταλήξουμε σε μια σύμφωνη γνώμη. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε. Βέμπερ, εκ μέρους των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Υπουργό για την παρουσίασή του. Θα είμαι σύντομη στα σχόλια και τις ερωτήσεις μου. Ουσιαστικά τρεις ερωτήσεις έχω. Μία για την Γενική Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ για την προστασία δεδομένων. Είπατε ότι σας ενδιαφέρει κάτι πιο φιλόδοξο. Θα ήθελα όμως να μου πείτε ακριβώς τι θέλετε να δείτε σε αυτή τη συμφωνία και πώς θα διασφαλίσετε ότι όσα επιτύχετε από τη συμφωνία αυτή θα εφαρμόζονται και για τις υπόλοιπες συμφωνίες που έχουν ήδη συναυθεί με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Δεύτερον, επανέρχομαι και εγώ στην Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας, το Investigation Order. Γνωρίζω από την εμπειρία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υπάρχουν τρομερά αποκλίνουσες απόψεις μεταξύ κρατών μελών. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη εμπιστοσύνης στα κράτη-μέλη όταν πρόκειται για θέματα της δικής τους αρμοδιότητας όπου τους ζητείτε να συνεργαστούν ή όπου δίνεται δυνατότητα σε άλλους να διεξάγουν έρευνες εντός του εδάφους τους. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πώς σκοπεύετε να προχωρήσετε προκειμένου να πετύχετε κάτι το ουσιαστικό για αυτό το θέμα της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας. Και εδώ περνάω και στον Ευρωπαίο Ισαγγελέα και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι θα μπει αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη της Προεδρίας της. μάλλον δεν ε, πιστεύω ότι μπορούμε και να επιτύχουμε κάτι εν πάση περιπτώσει. Επίσης αναφερθήκατε σε ένα σεμινάριο για την Eurojust που οργανώνεται το Σεπτέμβριο. Ως εισηγητήρια για τη Eurojust πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς δεν θα μπορέσω να παραβρεθώ γιατί όπως όλοι γνωρίζετε όταν κάτι συμπίπτει με την εβδομάδα της Ολυμέλειας στο Στρασβούργο συνήθως βρισκόμαστε όλοι στο Στρασβούργο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα είναι δύσκολο να διοργανώνετε κάτι και να περιμένετε να προσκαλέσετε μέλη του Κοινοβουλίου αν συμπίπτει με την εβδομάδα του Στρασβούργου. Ευχαριστώ. Επειδή έχουμε μακρύ κατάλογο μιλητών, θα ζητήσω από άλλους να κάνουν μία σύντομη ερώτηση ο καθένας και μετά θα ζητήσω από, τον Υπουργό να απαντήσει. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και πάλι συνεχίζοντας ε, με το θέμα της ερώτησης της συναδέλφου από την άλδε. Θα ήθελα να διατυπώσω την εξή ερώτηση. Η συμφωνία με τις ΗΠΑ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αν κατάλαβα καλά, υπάρχει μια προσέγγιση μεθοδολογική όσον αφορά ε, την εντολή που έχει προετοιμαστεί για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να ξέρω αν το Συμβούλιο ε, και πότε αυτή την εντολή θα την εγκρίνει και πότε θα μπορέσει αυτό να λειτουργήσει. Μπορείτε να μας πείτε μια προθεσμία μέχρι πότε ισχύει η διαρκή αυτή η προθεσμία πρέπει να είναι κανείς υπέρ μιας ε, δεσμευτικής ε, εντολής όταν πρόκειται για προστασία προσωπικών δεδομένων. Προστασία προσωπικών δεδομένων μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ΕΥΠΑ και συνεργασία μεταξύ δικαστικών αρχών και αστυνομικών αρχών και όταν ε, θα πρέπει εδώ να μην χάσουμε μια ευκαιρία και μία ερώτηση για τα προσωπικά δεδομένα και για τα δεδομένα των ταξιδιωτών στις σενάριες μεταφορές. Το Μάρτιο το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα για τα PNR, Passenger Name Records, τα όνα των ταξιδιωτών. Και πρόκειται για όλα τα στοιχεία των ε, ταξιδιωτών. Δεν είναι μόνο ένα θέμα δηλαδή σε σχέση με την ε, συμφωνία με τις ΗΠΑ. Θα πρέπει μέχρι τα μέσα Ιουλίου αυτό να μπορέσει να έχει ολοκληρωθεί. Καλείστε εσείς τώρα ως Βελγική Προεδρία να μπορέσετε να ε, μας πείτε κάτι γι' αυτό αν γίνεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σταβάρες και μετά Κλέης και μετά θα απαντήσει ο Υπουργός. Ευχαριστώ. Πολλές από τις ερωτήσεις που με ενδιαφέρουν έχουν ήδη γίνει και εμένα με ενδιαφέρει να ακούσω την άποψη του Συμβουλίου τόσο για το πλαίσιο προστασίας δεδομένων όσο και για τη, συμβασιση τη συμφωνία με συγχωρείτε PNR καθώς και για το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει για αυτές τις διαπραγματεύσεις και συμφωνίες. Συμφωνώ ότι τις προτεραιότητες της Βελικής Προεδρίας βλέπουμε την νόμιμη μετανάστευση. Πολλοί ευρωβουλευτές θεωρούμε ότι υπάρχουν πολλές κατασταλτικές διατάξεις για τη μετανάστευση πολλές από τις οποίες μπορεί και να μην είναι αποτελεσματικές, ενώ η βάση θα έπρεπε να είναι η νόμιμη μετανάστευση. Χαίρομαι λοιπόν που το βλέπω στην ημερήσια διάταξη της Προεδρίας, αλλά θα ήθελα να μου πείτε λίγο περισσότερα παραπάνω γι' αυτό. Και δύο σαφή ερωτήματα τώρα. Καταρχάς, ριζοσπαστικοποίηση. ακούγεται συχνά στην κοινή γνώμη, το βλέπουμε και στις εφημερίδες και στα blog, αλλά αυτή η έννοια της ριζοσπαστικοποίησης είναι υπερβολικά ευρία. Πολλοί που θεωρούν τους εαυτούς τους ριζοσπάστες δεν είναι βίαιοι τρομοκράτες εξτρεμιστές Άρα γιατί μιλάμε εδώ ακριβώς και επίσης το Συμβούλιο θα διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε διαδικασία παρακολούθησης αυτής της ριζοσπαστικοποίησης θα περνάει πρώτα από το Κοινοβούλιο για να έχουμε τον δημοκρατικό έλεγχο της διαδικασίας. Ένα άλλο θέμα τώρα. Επαναπατρισμός ε, προσφύγων. Αυτό το θέμα αφορά την επόμενη ακρόαση. Σας κόβω λοιπόν εδώ επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ωραία, σταματάω εδώ. Πολύ ωραία. Ο κύριος Κλέης και μετά θα απαντήσει ο Υπουργός. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι κύριε Υπουργέ, επισημάνατε και είπατε πιο πριν ότι η Βελγική Προεδρία θέλει να συνεισφέρει από πλευρά τη, ώστε να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή εισαγγελία. Και σύντομα, αν κατάλαβα καλά, θα διεξαχθούν συζητήσει στο Συμβούλιο. Θα διεξαχθούν, λέγω, ναι, συζητήσει στο Συμβούλιο και υπάρχουν αντίστοιχα μέτρα ακριβώς σε σχέση και με το ποινικό δίκαιο στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα να μου πείτε τι γίνεται συγκεκριμένα. Πώς ε, θα πάρει σάρκα και ωστά και θα λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Ποια είναι η πρόσθετη αξία που δημιουργείται και προσφέρεται από μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διότι έχουν εισαγγελίε στα κράτη-μέλη. Εδώ θα μπορούσε να υπάρξει μια βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και πώς θα γίνει σχετικά. Πρέπει να τεθεί το ερώτημα πώς μπορεί να δρά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από κοινού με τις Εθνικές Εισαγγελίες. Ευχαριστώ. Θα σας ζητήσω να απαντήσετε σύντομα στις ερωτήσεις που αφορούν τον τομέα σας και μετά θα περάσουμε στην επόμενη ακρόαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σύντομα, εν συντομία, κάποια στοιχεία να αναφέρω. Προστασία δεδομένων, προσωπικών δεδομένων. Φυσικά αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός ε, τομέας ως πεδίο. Και έγιναν και οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία SWIFT και έγινε και ε, η προσπάθεια καταπολέμησης και της τρομοκρατίας και υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό πρότυπο. Και είναι θέματα που μέσω διαπραγματεύσεων που ολοκληρώθηκαν ε, πρόσφατα και υπάρχει και διεξήχθη μια ευρύτερη συζήτηση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έγινε η προσπάθεια να δούμε πώς σε σχέση με τη ΣΥΠΑ ε, θα μπορέσει η Ευρώπη να σημειώσει πρόοδους. Οι συζητήσεις αυτές που έγιναν με τη ΣΥΠΑ ώστε να επιτευχθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων και μάλιστα προς όφελος των ευρωπαϊκών παραδόσεων σεβόμενοι τις ευρωπαϊκές παραδόσεις αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε μια δική μας μεθοδολογία και μέθοδο και πρέπει αυτή να μπορέσει να λειτουργήσει. Υπάρχουν διατάξεις ευρωπαϊκές και θα πρέπει αυτές στη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ να λειτουργήσουν. Και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να είναι μια σαφής προτεραιότητα που πρέπει να ισχύει για μας. Τούτου λεχθέντος φυσικά από την άλλη πλευρά δεν έχουμε φυσικά ολοκληρώσει ακόμα την πορεία μας. Δεν έχουν ολοκληρωθεί τα πράγματα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και διεξάγονται συζητήσεις από πλευρά του Συμβουλίου σε σχέση με μια τέτοια συμφωνία, ώστε να μπορέσει κατά τα τέλη του έτους να ε, ολοκληρωθεί το θέμα τη εντολής. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο ε, μπορεί να κλείσει υπό την Βελγική Προεδρία. Εμείς να προλιάνουμε το έδαφο μπορούμε μόνο. Και το θέμα της Eurojust, για παράδειγμα, και τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Λυπούμε που <clears throat> συμπίπτει από πλευρά ημερομηνία με την ε, χρονική εκείνη περίοδο που εσείς έχετε ανηλυμένες υποχρεώσεις και κολλείεστε. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και πρέπει να το ε, δούμε σε σχέση με τις διαβουλεύσεις. Πρόκειται για κάτι το οποίο θα βρει απήχηση και θα αντανακλάτε και στα έγγραφα τα οποία θα εξετάσετε εσείς ούτως ή άλλως στη συνέχεια. Αλλά δεν μπορούμε να ε, αν μείνουμε, ε, ώστε να υπάρξει ένα λεπτομερές ε, δρομολόγιο για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όταν θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις και οι διαβουλεύσεις για τη Eurojust θα πρέπει τότε να προβληματιστούμε και να δούμε πώς αυτή η συντονιστική δράση θα μπορέσει να εμβαθυνθεί σε σχέση με τον συντονισμό. Είμαι υπέρμαχος τέτοιου είδους θεσμών και θεσμικών πρωτοβουλειών και στο θέμα της διασυνοριακής του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει σε σχέση με τις εθνικές εισαγγελίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και με ποιο τρόπο μπορεί μια κοινή εισαγγελική αρχή να δράσει και να συντονίζεται. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί ώστε να καταλήξουμε και να δούμε ποιες δυνατότητες θα υπάρχουν στο μέλλον σε μια τέτοια Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Πιστεύω ότι κάποτε θα πρέπει να α, θα πούμε ότι χρειαζόμαστε αυτή την αρχή, αυτό το θεσμό. Βλέποντας πώς οι συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος διασυνοριακά δρούν και έχουμε προβλήματα εμείς να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτές τις δράσεις του οργανωμένου εγκλήματος, ε, τότε θα πρέπει να προωθηθούμε στο επίπεδο της εισαγγελική αρχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να μην παρακολιόμαστε. Υπάρχει ανάγκη για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ανταλλαγή απόψεων ώστε να οριμάσουν οι σκέψεις μας και να εμβαθύνουμε στις προτάσεις μας. Και έτσι νομίζω σε σχέση με την εντολή που αναφέρθηκα σχετικά ε, νομίζω ότι τα στοιχεία αυτά τα έχω ήδη καλύψει με την προηγούμενη τοποθέτησή μου και μετά σε σχέση με τους πρόσφυγες σίγουρα αυτό αφορά την αρμοδιότητα άλλου Υπουργού της Βελγικής Προεδρίας. Ευχαριστώ. Ε, επόμενη παρέμβαση πάλι στα Ολλανδικά. Σας ευχαριστώ και ε, καλωσορίζω την Βελγική Προεδρία και θέλω να πω ότι έχουμε υψηλές προσδοκίες ε, όσον αφορά την Βελγική Προεδρία και μπορώ να πω ότι η μέχρι τούδε Προεδρία βρισκόταν υπό την ε, συγκυρία της συνθήκης Λισαβόνας ούτως ή άλλως. Αναφέρθηκαν κάποια στοιχεία ώστε στην προηγούμενη, ας το πω έτσι, πρωτοβουλία, τα θεμελιώδη δικαιώματα διαδραματίζουν εδώ ένα πολύ σημαντικό ρόλο και το βρίσκω θετικό να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε σε αυτές τις πτυχές και να ασχοληθούμε με αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και όσον αφορά τώρα τις ε, ε, πτυχές η NPR, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σεπτέμβριο θα υποβάλει κάποια πρόταση, όμως θα έπρεπε να συζητήσουμε τις πτυχές αυτές και θα ήθελα να διατυπώσω την ερώτηση στο Συμβούλιο Κατά πόσον είσαστε πρόθυμοι να συνεργαστείτε με εμά ε, το Ευρωκοινοβούλιο. Είναι σημαντικό αυτό. Με το SWIFT είδαμε ότι είχαμε μεγαλύτερε δυσκολίε με το Συμβούλιο από ότι με του διατλαντικού μα φίλου Και έχει τεράστια σημασία τώρα εμεί στην Ευρώπη να μιλάμε με μία φωνή, να μιλάμε με μία ενιαία φωνή, εξεταζοντα τέτοια θέματα με τριτε χωρε Και δεν έχω υπόψη μου μόνο τις ΗΠΑ και τον Καναδά, αλλά και άλλε χώρε που μπορούν να προσθεθούν σε αυτόν τον κατάλογο π.χ. Σαουδική Αραβία, Κίνα και άλλες χώρες. Έχει τεράστια σημασία να έχουμε μια ευρωπαϊκή θέση ως τοποθέτηση, να μιλάμε με μια ευρωπαϊκή φωνή. Να μπορούμε σε σχέση με την εντολή, να μπορούμε ως κράτη-μέλη να έχουμε ενωμένε ε, μια ενιαία θέση. Τι γίνεται και σε σχέση με τις διμερείς συμφωνίες και το Visa Waiver Program. Για παράδειγμα το θέμα της α, ε, α, απαλλαγής διαβατηρίων τυπικών συγκεκριμένων χωρών με διμερείς συμφωνίες μεταξύ ΙΠΑ και των χωρών αυτών. Θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται ακριβώς και πώς μπορεί να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα και σε σχέση με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τι γίνεται, τι κάνετε εσείς και σε σχέση με την καταπολέμηση των απατών για παράδειγμα. Ξέρω ότι σε σχέση με το Βέλγιο θα ήθελα να μας πείτε τι κάνει η Βελγική Προεδρία. Λοιπόν, σύντομη ερώτηση, γιατί εδώ μιλήσαμε ήδη πολύ. Πριν από έξι μήνες, καλώς ορίζω βέβαια την Βελγική Προεδρία, αλλά πριν έξι μήνες έλεγα, ακούσαμε την Ισπανική Προεδρία που όρισε στόχους. Αλλά όλα δεν ευόδωσαν. Μετά από έξι μήνες έρχεται εδώ η Βελγική Προεδρία, η οποία οικιοποιείται τα ίδια, τους ίδιους στόχους ε, με τους, ε, με τους ίδιους όρους. Μιλήσαμε λοιπόν για την παιδοπορνογραφία, για την προστασία των ανηλίκων, για την καταπολέμηση της σωματεμπορίας. Λοιπόν, ρωτώ, σε έξι μήνες θα τελειώσει η Βελγική Προεδρία. Ποιος είναι ο στόχος ο οποίος είναι ο πρώτος πρώτος πρώτος στόχος των φιλοδοξιών σας. Λοιπόν, ποιος είναι ο πρώτος στόχος ε, μεταξύ όλων αυτών που αναφέρατε προηγουμένως. Ο κύριος Δίας Δεμέρα. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Λοιπόν, δύο πράγματα εμένα δεν μου φαίνονται καθαρά. Ρωτώ. Σχετικά με την εξαιρετική πρωτοβουλία των Ισπανών για, τον, για την Ευρωπαϊκή Τάξη Προστασίας, όλοι συμφωνήσανε στην ανάγκη να προστατεύσουμε τα θύματα. Μόνο κακοί άνθρωποι μπορεί να είναι αντίθετοι σε αυτό. Είπατε όμως και το σημείωσα ότι θα υπάρξει μια επαναδιατύπωση της Ισπανικής πρωτοβουλίας για τεχνικούς λόγους. Αυτό είπε και η κυρία Ρέντινγκ. Είπε δηλαδή ότι δεν διαφωνεί με την ουσία του ζητήματος αλλά οι διαφορές οφείλονται σε τεχνικές σε τεχνικά τερτύπια. Ρωτώ λοιπόν κύριε Υπουργέ, ποια είναι η κατάλληλη για σας νομική βάση και σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εμείς ακούσαμε την Σουηδική Προεδρία η οποία δεν είπε τίποτα, η Ισπανική Προεδρία είπε κάτι λίγο και τώρα ακούσαμε και εσάς που πάλι δεν λέτε τίποτα. Ξέρουμε ότι χρειάζονται 27 βουλήσεις ε, για να καταλήξουμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αλλά θέλω να ξέρω ποιες συγκεκριμένες δράσεις θα αναλάβει η Βελγική Προεδρία για να προωθήσει το θέμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Τι θα κάνει τελικά, θα γίνει αυτό το σεμινάριο το Σεπτέμβριο στην Μπρουζ όπου θα μπει και η εισαγγελία στο πακέτο Eurojust. Κυρία Βίγκστομ. Σας ευχαριστώ, ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε πώς εσείς ε, σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα σε σχέση με αυτή την συμφωνία μεταξύ ε, Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και την ενισχυμένη συνεργασία των κρατών μελών της Eurojust και της Europol. Πρέπει να πω ότι για, την, για μια κοινή θέση για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων που είναι σημαντική πτυχή είναι όμως και σημαντικό την άλλη πλευρά να θυμηθούμε ότι υπάρχουν ε, κάποια προβλήματα σε σχέση με τα κράτη-μέλη όσον αφορά τη στρατηγική. Το ακούσαμε και υπό την Σουηδική Προεδρία και υπό την ε, Ισπανική Προεδρία. Έχουμε και την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών που ακούστηκαν οι απόψεις τους σε σχέση με ε, την οδηγία, με την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν ώστε να είναι δυνατόν να διαμορφωθεί αυτό το πλαίσιο για το οποίο κάνουμε όλοι λόγο. Τώρα διαρωτώ με, η Βελγική Προεδρία δεν έχει μια εξαιρετική ας το πω έτσι προσέγγιση για να βελτιωθούν τα πράγματα όσον αφορά τα κράτη-μέλη. Και αυτό θα ήταν πολύ καλό, διότι όχι μόνο σε σχέση με το, τα κράτη-μέλη αλλά και για το ευρωπαϊκό επίπεδο και τα ευρωπαϊκά θεσμικά ε, όργανα είναι σημαντικό. Μια πολύ σύντομη ερώτηση, αν επιτρέπετε. Σε σχέση με τις ε, άτυπες συνεδριάσεις του Υπουργείου, αν βλέπω καλά τα πράγματα, την επόμενη εβδομάδα ή μάλλον όχι, ακόμα τούτη την εβδομάδα και δεν έχω τόσο μεγάλη πείρα από πλευράς προϋπηρεσίας ε, στην Ευρωβουλή αλλά σε σχέση με την άτυπη συνάντηση είναι σημαντική θέματα μακροπρόθεσμα για την λήψη αποφάσεων. Θα ήθελα να ξέρω ποια θέματα θα συζητήσετε στην επόμενη συνάντησή σας ώστε να γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται, ποια θέματα θα, επί ποιων θεμάτων θα διαβουλευτείτε. Ευχαριστώ. Δύο ακόμη σύντομε ερωτήσεις και μετά θα μπορέσετε να απαντήσετε. Η κυρία Αντζελίλη και μετά Μπαόρα. E Ευχαριστώ Υπουργέ. Με ικανοποίησε η αναφορά σας στην καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των ανηλίκων και την καταπολέμηση της παιδοπορνογραφίας. Θα ήθελα όμως να έχω μερικές πληροφορίες παραπάνω και για το χρόνο και για το περιεχόμενο για να μάθουμε δηλαδή αν αυτή η πρόταση αποτελεί όντως προτεραιότητα για τη Βελγική Προεδρία λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι αυτή η πρόταση έχει πολλαπλά συζητηθεί και η ομάδα μου το ΕΛΚ έχει οργανώσει ένα hearing στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ΛΥΜΠΕ στα τέλη Σεπτεμβρίου θα οργανώσει ένα hearing σχετικά. Λοιπόν, θα ήθελα να ξέρω παραπάνω. Ευχαριστώ. Μπάουερ. Η κυρία Έντιν Μπάουερ τώρα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπουργέ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για μια ανοιχτή ειλικρινή παρουσίαση και προσέγγιση από πλευρά της Προεδρίας για το θέμα της νέας οδηγίας για την καταπολέμηση του εμπορίου ανθρώπων της εμπορίας ανθρώπων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να σας ρωτήσω, να θέσω δύο ερωτήσεις. Όσον αφορά το σχέδιο αυτό το οποίο θα συζητηθεί και που εμπλέκεται η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Εμεί πήγαμε παραπέρα σε δύο πτυχέ σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ένα είναι το θέμα του Ευρωπαίου συντονιστή, διότι θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια ευρύτερη συνολική σφαιρική πολιτική ώστε να συντονίζονται οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές με μια ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή. Και το δεύτερο θέμα, οι κυρώσεις. Σε σχέση με τις κυρώσεις, εμείς προτείνουμε δίμευση και κατάσχεση των ε, ε, περιουσιακών στοιχείων τους, των ενόχων. Ποια είναι η άποψή σας για αυτές τις δύο πτυχές. Και η δεύτερη ερώτηση που θα ήθελα να θέσω είναι μεταξύ των θεμάτων που εσείς σκοπεύετε να εξετάσετε υπάρχει και ως θέμα η αναθεώρηση της οδηγίας σε σχέση με την προσωρινή άδεια ε, παραμονής διότι και αυτό αφορά το θέμα του, της εμπορίας ανθρώπων. Και, και αυτό συνδέεται και όλας άμεσα και με την προστασία των θυμάτων βίας και κακοποίησης. Ιντάργο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πέρα από τα καλωσόριζες, τα συνηθισμένα, να σας πω ότι με απαγοητεύσατε πλήρως διότι όταν μιλάτε εσείς για την ευρωτάξη και την προστασία των ε, γυναικών ε, εσείς αρχίζετε και λέτε διάφορα για το οργανωμένο έγκλημα και τη βία που ασκεί στις γυναίκες. Μα εσείς όμως είστε προεδρεύον και προσωπείτε μια δημοκρατική χώρα. Δεν μπορείτε να λέτε τέτοια πράγματα. Και θέλετε να τα έχετε και καλά με την κυρία Ρέντινγκ και όλα τα σχετικά. Αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σκέφτεται η κυρία Ρέντινγκ για αυτό το θέμα. Μα η κυρία Ρέντινγκ δεν έχει κανένα πρόβλημα να κυκλοφορεί ένα της Ευρώπας. Εκείνες που πραγματικά απειλούνται είναι εκείνες οι γυναίκες που τις κυνηγάνε οι πρώην και δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν και να πάνε πουθενά. Όχι φυσικά η κυρία Ρέντινγκ. Λοιπόν ή θα το πάρετε σοβαρά το θέμα ή αλλιώς θα είστε μία θρασίδηλη προεδρία. Αναλάβετε το λοιπόν το θέμα με πραγματική ευθύνη και αναλάβετε και τις ευθύνες σας για να προστατεύσετε τις Ευρωπαίες γυναίκες και όχι να το γυρνάτε το θέμα σε μια γενικόλογη συζήτηση οργανωμένου εγκλήματος. Ευχαριστώ. Ζητάμε από τον Υπουργό να μας απαντήσει. Όπως βλέπετε πρόκειται για πολλά θέματα δύσκολα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολλές ερωτήσεις βέβαια διατυπώθηκαν. Δεν έχουμε την δυνατότητα τώρα εδώ κατά λεπτός εξειδικευμένα να τις απαντήσω. Αλλά δεν πρέπει να ακολουθούμε κάποια απλά, απλοϊκά, ας το πω έτσι, σχήματα ε, τύποποιημένη σκέψη. Εμείς θέλουμε το ένταλμα προστασίας όπως ξεκίνησε από την Ισπανική Προεδρία να το συνεχίσουμε. Θέλουμε να ολοκληρωθεί και θέλουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να σημειωθούν πρόοδοι. Και τα προβλήματα αυτά ε, της βίας εις βάρος των γυναικών να αντιμετωπιστούν. Αυτή είναι μία πτυχή. Φυσικά υπάρχουν και άλλες πτυχές, έτσι δεν είναι παράδειγμα η εμπορία ανθρώπων. Και εδώ φυσικά πρέπει να κάνουμε πάλι ό,τι περνάει από το χέρι μας, να προστατέψουμε τις γυναίκες από κάθε μορφή βίας. Να απαντήσω πρώτα σε μία ερώτηση που μου διατυπώθηκε. Δηλαδή, ποιες είναι οι φιλοδοξίες της Προεδρίας. Θα ήθελα εδώ ταπεινά να εκφραστώ. Εξάμεινη είναι η Προεδρία μας, έτσι. Εξάμεινη Προεδρία και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιομορφία του Βελγίου στην πολιτική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Βέλγιο, θέλουμε να κάνουμε πραγματικά ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε με την Προεδρία μας που θα εργάζεται 200% και όχι 100% γνωρίζουμε ότι υπάρχουν περιορισμοί και ότι δεν μπορούμε όλα να τα πετύχουμε. Υπάρχει η εναλλασσόμενη Προεδρία και πρέπει κάποια πράγματα να μπορέσουν να προσαρμοστούν, να τα ξεκινήσουμε, να τα συνεχίσουμε και να προσαρμοστούν. Πρέπει αυτή η συνέχεια και η συνεκτικότητα να διασφαλιστεί. Νέος προβληματισμός να υπάρξει, νέες εταιρικές σχέσεις να δημιουργηθούν. Όταν με ρωτάτε ποιες είναι οι φιλοδοξίες μου, ε, τότε πρέπει να απαντήσω ότι εμείς, εγώ, εμείς στο Βέλγιο, στην Ευρώπη, θέλουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα, να βελτιώσουμε την Ευρώπη, να βελτιωθεί η Ευρώπη στη λειτουργία της στους πιο διαφορετικούς τομείς στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν κάποιες πτυχές που προανέφερα και που είναι σημαντικές. Όμως από την άλλη πλευρά πρέπει να πετύχουμε μεθοδολογικά να βρούμε τη σωστή προσέγγιση, ώστε τα αποτελέσματα να βελτιωθούν. Με κάθε ταπεινοφροσύνη θα γνωρίζω ότι το ένα ή το άλλο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κάποιες ατέλειες, κάποιες, ε, ε, κάποιους περιορισμούς. Παρόλα αυτά όμως πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες να καταλήξουμε σε θετικά αποτελέσματα. Για τα θεμελιώδη δικαιώματα είπε κάποιος ότι δεν έχω πει τίποτα, όμως θα ήθελα να πω ότι υπάρχει εδώ φυσικά και το θέμα των συμφωνιών για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύμβαση, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επίσης αναφέρθηκα και στην δυνατότητα να μπορούν οι άνθρωποι καλύτερα να προστατεύονται. Είναι πολύ συγκεκριμένες λοιπόν χειροπιαστές πρωτοβουλίες αυτές που τίθενται στο τραπέζι και που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Διατυπώθηκε μια ερώτηση επίσης για τα δεδομένα των ταξιδιωτών στις εναέριες μεταφορές των επιβατών ε, των αεροπλάνων. Θα αναμείνουμε το Σεπτέμβριο και την πρωτοβουλία και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα δεν γνωρίζω γιατί αναφέρθηκε το θέμα προβλημάτων με το Συμβούλιο. Δεν έχω μακρά πείρα βέβαια, αλλά έχω το βίωμα, την πείρα, ότι στο Συμβούλιο Υπάρχει φιλόδοξη προσπάθεια να ρυθμιστούν και να διευθετηθούν κάποια θέματα με θετικό τρόπο και στο Συμβούλιο νομίζω και με το θέμα SWIFT υπήρξε σωστή αντίδραση και έτσι σωστά υπήρξε η δραστηριοποίηση από πλευράς μας. Τώρα, σε σχέση με ελέγχους όσον αφορά ε, κάποια θέματα, αυτό είναι βέβαια οπωσδήποτε προτεραιότητα δική μας να υλοποιηθούν αυτές οι προτάσεις. Και αυτό το οποίο αναφέρθηκε σε σχέση με την, το ένταλμα προστασίας, πώς θα μπορέσει να προσαρμοστεί εδώ επιτρέψτε μου να, αναφερθώ στην ε, συζήτηση επί των θεμάτων αρχής ε, που προηγήθηκε. Τα θύματα λοιπόν πρέπει να προστατεύονται και στη χώρα εκείνη στην οποία έχουν την κατοικία τους και την έδρα τους, ας το αποκαλέσω έτσι. Υπάρχουν διαφορετικές νομικές ε, ε, διατάξεις. Πρέπει να διαφοροποιήσουμε τα πράγματα μεταξύ ποινική δικονομίας και ε, ποινικού δικαίου και αστικού δικαίου. Πρέπει να δούμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Εδώ η συζήτηση είναι όμως σαφής. Υπάρχει νομική βάση και μέσα στο πλαίσιο του Συμβουλίου θα θέλαμε άμεσα, βραχυπρόθεσμα, άμεσα να σημειωθούν πρόοδοι. Τώρα, για το θέμα της Ευρωπαϊκής μου ζητήσατε και με ρωτήσατε συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις. Επαναλαμβάνω, σε ένα σεμινάριο για τη Eurojust θα συζητηθούν αυτά και στο άτυπο συμβούλιο αυτή την εβδομάδα πάλι ακόμα. Δεν θα υπάρξει ε, η, η διευθέτηση, η ίδρυση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε αυτό το επίπεδο, σε αυτή τη φάση. Θέλουμε να υπάρξει ένα κοινοτικό μέσο το οποίο θα αναπτυχθεί περαιτέρω. Η Eurojust είναι ένα σημαντικό βήμα και η συνάντηση όλων των εισαγγελέων και των εισαγγελικών αρχών είναι ένα περαιτέρω βήμα ώστε η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των εισαγγελικών αρχών να βελτιστοποιηθεί. Ένα άλλο βήμα είναι μια εισαγγελική αρχή που θα είναι ομοσπονδιακού χαρακτήρα. Είμαι υπέρμαχος εγώ και πιστεύω ότι θα γίνει αυτό ε, μακροπρόθεσμα. Δεν υπάρχει όμως κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία ώστε μέχρι τα τέλη του έτους ε, να ευδοκιμήσει αυτός ο στόχος. Θα πρέπει να προβληματιστούμε για αποτελεσματικές μεθόδους για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και να προβληματιστούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα ε, κακοποίηση παιδιών και χρήση του διαδικτύου σε σχέση και με κακοποίηση των παιδιών. Είπα ότι το θέμα της κακοποίησης παιδιών τίθεται και στο διαδίκτυο. Υπάρχει μια σειρά πρωτοβουλειών σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να σκεφτούμε τώρα πώς οι πρωτοβουλίες θα εναρμονιστούν ώστε αυτή η κακοποίηση μέσω, ή τα θέματα τα οποία οδηγούν σε κακοποίηση μέσω του διαδικτύου να καταπολεμηθούν ως συνιστώσεις. Πώς είναι δυνατόν για παράδειγμα να είναι ποινικέ οι πράξεις αυτές από πλευρά ενηλίκων που εμπλέκονται σε σχέση με το διαδίκτυο σε θέματα κακοποίηση παιδιών και χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ε, ώστε να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς τους. Αυτό πρέπει να δούμε και να μπορέσουμε αποτελεσματικά να καταπολεμήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να δημιουργήσουμε κέντρα για την καταπολέμηση αυτή τη εγκληματικότητα, να προστατευτούν τα θύματα, ιδιαίτερα ανήλικοι και παιδιά. Και εδώ συγκεκριμένα μέτρα θα πρέπει πρέπει να εναρμονιστούν για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Θα λέγα κυρία Πρόεδρε, με αυτά τα οποία είπα, ότι σε πολλά σημεία μπόρεσα να δώσω μια απάντηση επαρκώς. Πολλές πτυχές αναφέρθηκαν και επανειλημμένα ε, τέθηκαν κάποια θέματα. Αν ξέχασα κάτι να μου το αναφέρετε για να επανέλθω. Ελπίζω όμως ότι και σύντομα θα έχουμε τη δυνατότητα να προβούμε σε μια συγκεκριμένη ανταλλαγή απόψεων και πάλι. Ευχαριστώ. Μπορούμε να συνεχίσουμε την συζήτηση. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τώρα με τα θέματα εσωτερικών υποθέσεων και τις εκεί προτεραιότητες της Βελγικής Προεδρίας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας στη συνεδρίασή μας. Θα ήθελα να υποδεχθώ την Υπουργό Ανεμή Τεμπού και θα συνεχίσουμε με τις προτεραιότητες της Βελγικής Προεδρίας σε θέματα εσωτερικών υποθέσεων, ασφάλειας κτλ. Πρόκειται για θέματα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Επιτροπή μας. Έχετε το λόγο για να κάνετε την εισαγωγή σας και μετά θα ακούσουμε διάφορες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να σας μιλήσω για τις προτεραιότητες της Βελγικής Προεδρίας και τα θέματα εσωτερικών. και φυσικά δεν θα μακρηγορήσω ιδιαίτερα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε μετά κύριοι βουλευτές. Θα ξεκινήσω με τη συνθήκη της Λισαβόνας όπου πλέον βρισκόμαστε σε θέση ισοτιμίας και μπορούμε να συγκρίνουμε τις αρμοδιότητές σας με αυτές του Αμερικανικού Κογκρέσου. Υπάρχει λοιπόν ισοτιμία και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση που έχουμε σήμερα στο Κοινοβούλιο. Διότι τα τρία θεσμικά όργανα πρέπει να συνεργαστούμε. Το Βέλγιο ήταν πάντα μια ιδιαίτερα προευρωπαϊκή χώρα που θέλει να καλύψει το ρόλο του κατά την Προεδρία αλλά και να σεβαστεί και τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τη Λισαβόνα. Σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο θέλουμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα στον τομέα της ασφάλειας. Η Ισπανία έχει ξεκινήσει ένα, ένα σχέδιο για την ασφάλεια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ορισμένες μορφές εγκληματικότητας που μπορούν να καταπολεμηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ισπανική Προεδρία έκανε τα πρώτα βήματα Εμείς σίγουρα δεν θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας, αλλά θέλουμε τουλάχιστον να διαμορφώσουμε τη μεθοδολογία αυτού του συστήματος και ο προκάτοχός μου, ο Ισπανός ε, συνάδελφος, ήδη έχει ορίσει τα όρια αυτής της μεθοδολογίας και εμείς μετά θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αναλύσουμε τις πληροφορίες, να ανταλλάξουμε πληροφορίες για να έχουμε μία σαφή ανάλυση των εγκληματικών φαινομένων στην Ευρώπη. θα μπορέσουμε πιστεύω ούτως να ορίσουμε τις προτεραιότητες γιατί στον τομέα της δικαιοσύνης χρειάζονται οι αποφάσεις γιατί μέσα από τις αποφάσεις μόνο μπορούμε να έχουμε και συγκεκριμένα μέτρα. Το σχέδιο Harmony κατά την Προεδρία μας θα είναι πολύ σημαντικό. Πρόκειται για ένα κοινό σχέδιο μεταξύ Προεδρίας και Κομισιόν και στα τέλη της χρονιάς φέτος θα έχουμε και τον πρώτο απολογισμό. Και η Επιτροπή Εσωτερικών θα πρέπει και αυτή να εκπληρώσει τον, το ρόλο της. Η λειτουργική πλευρά είναι πολύ σημαντική. Εάν μέχρι τα τέλη του 2010 θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία για τα θέματα της ασφάλειας, τότε μέχρι το 2014 θα έχουμε μία αποτελεσματική στρατηγική εσωτερική της δικαιοσύνης που ελπίζουμε ότι θα είναι και λειτουργική. Αυτά όλα θα γίνουν και βάσει των πληροφοριών που θα έχουμε θέλουμε εμείς πάντα να έχουμε μία σφαιρική τοποθέτηση και έχουμε αναλάβει στοχευμένες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήδη σήμερα έχουμε μερικά διεθνικά φαινόμενα. Ξέρουμε ότι η εγκληματικότητα δεν σταματάει στα εσωτερικά σύνορα. Έχουμε λοιπόν, είπαμε, διεθνικά φαινόμενα τα οποία θα πρέπει να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε. Δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Χρήση, παράνομη χρήση όπλων. Η χρήση αυτών των όπλων αυξάνεται όχι για πολεμικούς λόγους αλλά για εγκληματικούς λόγους. Δηλαδή για ληστείες. Ζήτησα λοιπόν από την Ευρωπόλ να μας δώσουν οδηγίες, να μας πούν τι κάνουν για να απαγορευτούν τα όπλα. Είπαμε δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει πρόληψη. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πώς κυκλοφορούν όλα αυτά τα όπλα στην Ευρώπη και εμείς βάση της έκθεσης Europol θέλουμε να εξετάσουμε, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του, να καταλάβουμε ποια είναι τα απαραίτητα μέσα που μπορούμε να αξιοποιήσουμε ας πούμε μια οδηγία για να μπορέσουμε να συντονίσουμε τις δράσεις μας χρειάζεται περισσότερη πληροφόρηση, περισσότερες ανταλλαγές. Πρέπει να βρούμε λοιπόν μια μεθοδολογία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το λαθρεμπόριο όπλων. Επίσης, ένα άλλο βασικό πρόβλημα. Η οδική ασφάλεια, καθημερινή βία, με στο σπίτι. Πώς μπορούμε για να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά, να έχουμε μία ευρωπαϊκή άποψη. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε ένα διάλογο βασισμένο στις εμπειρίες όλων των κρατών μελών Και αυτή θα είναι μια άλλη προτεραιότητα της Προεδρίας μας. Για... Πέρα από αυτά τα δύο βασικά σημεία, ανταλλάσσοντας πληροφορίες μπορούμε να ενημερωνόμαστε για το πώς καταπολεμούνται αυτά τα φαινόμενα στα άλλα κράτη-μέλη. Και ένα άλλο πρόβλημα είναι η πρόληψη του ριζοσπαστισμού, του βίαιου ριζοσπαστισμού. Γι' αυτό λοιπόν κατά την προεδρία μας θα ξεκινήσουμε το σχέδιο κόμπρα και θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε μέσα στα πλαίσια του σχεδίου όλες τις ανταλλαγές πληροφόρησης. Θέλουμε να έχουμε πρόληψη για αυτά τα βία ριζοσπαστικά φαινόμενα. Θα Θέλουμε να φτιάξουμε και ένα εγχειρίδιο, έναν οδηγό για τους αστυνομικούς. Θέλουμε να εκπαιδεύσουμε την κοινωνία να επαγρυπνεί για πρωτοβουλίες κατά της τρομοκρατίας. Θέλουμε λοιπόν ως Βελγική Προεδρία να αναλυφθούν Πρωτοβουλίε στον τομέα αυτό. Ένα άλλο ζήτημα είναι το ΣΥΣ 2. στο Συμβούλιο της 5ης και 6ης Οκτωβρίου θέλουμε να ορίσουμε ένα χρονοδιάγραμμα και να έχουμε ένα συγκεκριμένο απολογισμό για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Όταν μιλάω για λαθρεμπόριο όπλων, για εγκληματικότητα στο δρόμο, είναι σημαντικό να ξέρουμε πώς θα ανταλλάσσουμε πληροφορίες. Το ΣΥΣ 2 είναι ένα ουσιαστικότατο σχέδιο. Πρέπει λοιπόν εμείς να εγγυθούμε το σύστημα να είναι αποτελεσματικό, να ξεκινήσει εγκαίρως. Οπότε θα είναι πολύ σημαντικό το τι θα, κάνει, θα πει το Συμβούλιο. Υπάρχει και συζήτηση για τον οργανισμό για την IT. Θα πρέπει να αποφασίσουμε πού θα είναι η έδρα αυτού του οργάνου και πώς θα λειτουργεί. Και φυσικά οι αρμοδιότητες θα πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο. Λοιπόν κυρία Πρόεδρε, εγώ δεν ήθελα να ξεκινήσω με έναν κατάλογο 500 και πάνω μέτρων που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ήθελα απλώς να σας δώσω μια συνοπτική ιδέα για το τι θα κάνουμε υπό Ισπανική είπαμε Προεδρία, είμαστε μια προευρωπαϊκή χώρα. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια προευρωπαϊκή προοπτική για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα υπάρχοντα προβλήματα στα κράτη-μέλη και να ορίσουμε δύο-τρεις προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια. Στόχος μας είναι μέχρι το 2014 να μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια πολιτική, κοινή πολιτική εσωτερικών ούτως ώστε τα τρία όργανα να μπορούν να εργαστούν για ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας, για να έχουμε μια Ευρώπη πιο ασφαλή. Σας ευχαριστώ. Θέσατε κάποια θέματα για τα οποία είχαμε ρωτήσει και προηγουμένως, όπως για παράδειγμα η ριζοσπαστικοποίηση. Θα ζητήσω πρώτα από τους συντονιστές να κάνουν ερωτήσεις και να απαντήσετε. Μας πιέζει και ο χρόνος και μετά θα ακούσουμε και τα υπόλοιπα μέλη. Ο κύριος Μπουσουτείλα, εκ μέρους ε, των συντονιστών. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, μιλώ εκ μέρους ε, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αναφερθήκατε αρκετές φορές στην κόση. Μία ανησυχία δική μου, παρόλο που μας ενδιαφέρει τρομακτικά αυτή η Επιτροπή, είναι ότι δεν μας αφήνει την εντύπωση αυτή η Επιτροπή ότι βρίσκεται υπό κοινοβουλευτικό έλεγχο, υπό οποιονδήποτε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και αυτό το σημείο θα ήθελα να το σημειώσω, γιατί παρά τη σημασία αυτής της Επιτροπής και της αρμοδιότητάς της που είναι ιδιαίτερη σημασία και για την Επιτροπή μας δεν βλέπω να υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος. Τώρα, κάποια πράγματα ακόμη όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Ως εισηγητής για το Frontex, ένα πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι η επεξεργασία δεδομένων από το Frontex. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει προτείνει κάτι τέτοιο παρόλο που αρχικά υπήρχε ενδιαφέρον για να δοθεί τέτοια αρμοδιότητα στην υπηρεσία Frontex και γνωρίζω ότι αυτό το θέμα έχει συζητηθεί αρκετά στο Συμβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την άποψη της Προεδρίας σχετικά. Τέλος, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό TFTP, τι. Γνωρίζετε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την ψηφοφορία για το SWIFT. Είναι στόχος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης των τρομοκρατών. Τι θα κάνει το Βέλγιο για να περάσει αυτό όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στη Βαρόνι Λάτφορντ εκ μέρου των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ. Μου ζήτησε ε, ο συνάδελφος να μιλήσω εκ μέρους της ομάδας. Σας ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ. Χαιρόμαστε που ακούσαμε τις προτεραιότητές σας όσον αφορά την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος των διεθνών συμμοριών. Συχνά μένουμε με την εντύπωση ότι δεν έχει αποδοθεί απαραίτητη σημασία σε αυτό το θέμα την τελευταία δεκαετία, σε σύγκριση για παράδειγμα με την τρομοκρατία. Επίσης, ποια είναι η άποψή σας όσον αφορά θέματα όπως ε, το παράνομο εμπόριο όπλων. Πέρα από αυτό τώρα, καταρχάς όπως ε, και ο κύριος Μπουσουτήλ με ενδιαφέρει να ακούσω τι έλεγχο θα έχουμε στην Επιτροπή Κόζη. Όμως πέρα από αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες ακριβώς είναι οι προθέσεις σας για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης. Θα ήθελα όμως να σας κάνω έκκληση να εγκαταλείψουμε αυτόν τον όρο. Το να είναι κάποιος ριζοσπάστης δεν σημαίνει ότι έχει σχέσεις με την τρομοκρατία. Όταν κάποιος είναι φονταμενταλιστής, επίσης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι εξτρεμιστής ή τρομοκράτης. Θεωρώ ότι αυτός ο όρος, ριζοσπάστης, δεν είναι χρήσιμος στην περίπτωσή μας. Και όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για εντοπισμένους ριζοσπάστες, φαίνεται ότι σκοπεύει να καλύψει και όλους τους διαφωνούντες, τους διαμαρτυρόμενους σε οποιονδήποτε τομέα. Νομίζω ότι αυτή είναι μια επικίνδυνη πορεία. Αν οποιονδήποτε διαμαρτύρεται, τον εντοπίζουμε ως ύποπτο τρομοκρατίας. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει πολύ σαφής διαχωρισμός. Και επίσης θα ήθελα να ζητήσω από τη Βελική Προεδρία να περάσει καλύτερα στην προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Εντάλματος ε, Σύλληψης και να ζητήσω και τη συνεργασία των κρατών μελών σχετικά γιατί αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι σε άσχημη φάση. Σαντζετίνη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν πρώτα θα ήθελα να προσυπογράψω τα επιχειρήματα της Βαρόνης Λάτφορντ το ότι ο φονταμενταλισμός είναι κάτι τελείως διαφορετικό σε σχέση με την απειλή και ότι εδώ η διατύπωση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό υποστηρίζω απόλυτα αυτά τα οποία προανέφερε στην παρέμβασή της. Προσέξτε, είπατε ότι θα θέλατε να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα και το οργανωμένο έγκλημα αμέσως ανήκει σε αυτό το θέμα των ναρκωτικών και το εμπόριο ναρκωτικών δεν έχω υπόψη φυσικά φάρμακα, αλλά σκληρά ναρκωτικά και οπιούχα. Και θα ήθελα να μου πείτε αν μέσα στο πλαίσιο της καταπολέμησης της, της ε, του οργανωμένου εγκλήματος ασχολείστε και με αυτό, διότι αυτό έχει δύο πτυχές, δύο όψεις του νομίσματος φυσικά υπάρχουν. Κάθε έχει την αίσθηση ότι αν είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί στην καταπολέμηση κάποτε θα επιληθεί το ζήτημα, αλλά φαίνεται ότι οι επιτυχίες δεν είναι δεδομένες. Από την άλλη πλευρά, υπό ένα άλλο πρίσμα μπορεί να ασχοληθεί κανείς με τα ναρκωτικά, υπό το κοινωνικό πρίσμα δηλαδή. Όταν πρόκειται για διασύνορια κακά διοργανωμένο οργανωμένο έγκλημα διαρωτώ με πού βρίσκεστε, πού, πώς τοποθετήστε όταν πρόκειται για εμπόριο ναρκωτικών. Και μια τελευταία συγκεκριμένη ερώτηση αφορά την ε, υπηρεσία ή e τι. Είπατε τους επόμενους έξι μήνες θα θέλατε να ολοκληρώσετε να ληφθεί μια απόφαση σχετικά. Η ειπατε τους επομενους εξι μηνες θα θελατε να ολοκληρωσετε να ληφθει μια αποφαση σχετικα η γαλλια και η Εσθονία έχουν προβλήματα σε σχέση με αυτό. Και διαρωτώ με, θα μπορούσατε τώρα να μας πείτε ίσως πώς έχουν τα πράγματα, πώς έχουν προχωρήσει αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ταβάρες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ μια ερώτηση για την ριζοσπαστικοποίηση. Και ήθελα τόσο πολύ να κάνω αυτή την ερώτηση που την έκανα και πριν στον Υπουργό δικαιοσύνη. Εν πάση περιπτώσει, ουσιαστικά συμβαδίζω με τη Βαρόνη Λάτφορντ. Καταλαβαίνουμε τι βρίσκεται πίσω από την ανησυχία για τη ριζοσπαστικοποίηση. Δηλαδή το να προσπαθήσουμε να βρούμε τα αίτια της τρομοκρατίας. Και μέχρι εκεί ακούγεται θέμα με καλές προθέσεις. Όμως έτσι μπαίνουμε στον αγώνα των ιδεών και δυστυχώς ε, το Συμβούλιο δεν είχε ασχοληθεί με το θέμα αυτό από την αρχή. Όμως αυτή τη στιγμή το έγγραφο είναι τόσο ευρύ που θα μπορούσε να συμπεριλάβει όλους τους ριζοσπάστες βίους ε, και μη και σίγουρα πρέπει να θυμάστε ότι υπάρχουν και πολλοί από εμάς που γινόμαστε ριζοσπάστες και είμαστε περήφανοι για αυτό. Άρα λοιπόν κάτι τέτοιο αν περάσει στην κοινή γνώμη δεν θα είναι καθόλου χρήσιμο. Επομένως, αν θέλει να ξεκινήσει καλά το Συμβούλιο, μια καλή λύση θα ήταν να ξεκινήσετε από το Κοινοβούλιο που είναι ανοιχτό στην κοινωνία των πολιτών και όπου μπορεί να υπάρξει καλός έλεγχος και συζήτηση τέτοιων προτάσεων γιατί αυτός ο μυστικοπαθής τρόπος πορείας θα δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον. Περισσότερο σχόλιο παρά ερώτηση έκανα. Εν πάση περιπτώσει θέλω να ρωτήσω ακριβώς τι εννοείται όταν μιλάτε για τη μετώπιση της ριζοσπαστικοποίηση. Έκτος και μετά θα απαντήσει η υπουργό στις πρώτες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Υπουργέ, Εσείς αναφερθήκατε στην καταπολέμηση της θρηζοσπαστικοποίησης και είπατε ότι η Βελγική Προεδρία θα ήθελε να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Είναι σημασιολογικές ίσως ε, οι διαφοροποιήσεις. Τι εννοούμε ακριβώς, την Ισλαμοποίηση, τον Ισλαμικό φονταμενταλισμό, ίσως αυτό θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το Βέλγιο εδώ είναι μια επιμελητιακή πλατφόρμα θα έλεγα υποστήριξης ή τέλος πάντων παροχής πολλές φορές συνδρομής σε Ισλαμιστές ε, δράστες όπως για παράδειγμα σε σχέση με τον Μασούντ και το πλήγμα της Αλκάιντα στη Μαδρίτη ε, τα ίχνη ε, εντοπιζόντουσαν μέχρι και το Βέλγιο και γι' αυτό λοιπόν η Βελγική Προεδρία ακριβώς κατά της Ισλαμικής ακραίας αυτής ριζοσπαστικοποίησης θα έπρεπε να δράσει. Τι εννοείται όμως ακριβώς προληπτική δράση. Είσαστε υπέρμαχος μιας αυστηρής ε, κυρωτικής θα έλεγα καταστολής δράσης έναντι των ε, ενόχων. Ε, θα πρέπει να το δούμε αυτό ότι υπάρχουν κάποιοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίοι απευθύνουν έκκληση να υπάρξει χρήση βίας. Υπάρχει επίσης ε, λογοκρισία. Εδώ τι είναι ριζοσπαστικοποίηση για σας. Ποια είναι τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιείτε σε σχέση για παράδειγμα με την ελεύθερη έκφραση των πολιτών. Θα θέλατε κατασταλτικά μέτρα να ληφθούν, ιδιαίτερα όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, ιδιαίτερα όσον αφορά την Ισλαμική αυτή τοποθέτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ζητήσω από την Υπουργό να απαντήσει μέχρι στιγμής και μετά θα συνεχίσουμε με δεύτερο γύρο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω σύντομα να απαντήσω στις ερωτήσεις που διατυπώθηκαν. Πρώτα απ' όλα καταρχήν για την υπηρεσία IT. IT. Δεν μπορώ να πω τίποτα αυτή τη στιγμή για αυτήν. Σίγουρα μια σειρά επαφών και συζητήσεων θα προηγηθούν και σε σχέση με τους επόμενους μήνες σίγουρα κάποιες αποφάσεις ε, ε, θα μπορούσαν να ληφθούν. Τους επόμενους όμως έξι μήνες υπό την Βελγική Προεδρία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτές τις πτυχές. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι χρειαζόμαστε αυτό τον οργανισμό, αυτή την υπηρεσία IT, IT e την χρειαζόμαστε. Το θέμα της έδρας θα πρέπει να το αποσαφηνίσουμε, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσει να αρχίσει να λειτουργεί αυτή η υπηρεσία και αν δεν καθορίζαμε την έδρα της θα ήταν αρνητικό. Και εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο τους επόμενους μήνες θα πρέπει να υπάρξουν μέρημνες ώστε ο προβληματισμός να ευδοκιμήσει. Τώρα το θέμα των ναρκωτικών που προαναφέρθηκε και το θέμα των, των, θέμα των όπλων ε, Έχω υπόψη εδώ την, το σύμφωνο, το γαλλικό σύμφωνο κατά των ναρκωτικών. Περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται σίγουρα για μία από τις προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν ε, αντίστοιχοι φορείς ε, και θεσμικά όργανα που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Για μένα όμως είναι πολύ σημαντικό να δούμε σε ποια πλευρά βρισκόμαστε και σε σχέση με τις συμμορίες, ε, μετακινούμενες συμμορίες και το θέμα των όπλων, των πυροβόλων όπλων είναι σημαντικό. Είναι και θέμα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Να βοηθάει το ένα κράτος το άλλο, ώστε οι ροές των ναρκωτικών να αποκαλυφθούν, να δούμε πώς διακινούνται τα ναρκωτικά και το πρόβλημα να το χτυπήσουμε στη ρίζα του. Ουσιαστικά πρόκειται για θέμα αρχής που είναι το ίδιο φαινόμενο και για τα πυροβόλα όπλα και για τα όπλα και για τα ναρκωτικά. Χρειαζόμαστε περισσότερο περισσότερες πληροφορίες, ανταλλαγή πληροφοριών και καλύτερη συνεργασία, βελτιωμένη συνεργασία. Τήθηκε, τέθηκε το ερώτημα για την κόζη. Αν δεν κάνω λάθος, από τον κύριο Κούκερμπεργκ, τον Γενικό Γραμματέα της κόζη που θα προσέλθει, ε, θα υπάρξει πληροφόρηση. Γνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν εντάσσεται το θέμα στο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Υπάρχει μια νέα δομή, μια νέα δομή και πρέπει τα πράγματα να μετεξελιχθούν και η πρακτική να ε, μετεξελιχθεί καλύτερα. Για μένα βρίσκονται αυτά όλα σε μετεξέλιξη εν ροή, εν ρευστό. Για το, την κόση περί τίνος πρόκειται πώς η κόση πραγματικά θα προετοιμάζει, θα προλυαίνει το έδαφος στο πολιτικό επίπεδο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε σε συγκεκριμένο νομοθετικό έργο να μπορεί να υπάρχει, να διασφαλίζεται η ανταλλαγή πληροφοριών και να διασφαλίζεται η σωστή βάση πληροφόρησης. Και σε σχέση τώρα με το TFTP, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, πρέπει να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ. Για το SWIFT πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για έναν τομέα που αφορά την δικαστική συνεργασία, θέματα δικαιοσύνης. Και εδώ τίθενται και τα θέματα των αρμοδιοτήτων στο δικαστικό επίπεδο. Για την Frontex ίσως είναι πιο απομονωμένη η θέση του Βελγίου. Εμείς δεν είμαστε υπέρ του αυτά τα στοιχεία να τα επεξεργάζονται ή της Frontex και εκείνοι να τα διαχέουν. Τώρα, από κοινού, σε σχέση με το ΣΥΣ Schengen Information System, όχι, διορθώνει η Υπουργό. Πρόκειται για το θέμα της ριζοσπαστικοποίησης και της καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης. Η καλύτερη μέθοδος είναι η πρόληψη, η πρόνοια. Έτσι μπορούμε να μεριμνήσουμε να καταπολεμηθούν το δυνατόν πιο γοργά ε, οι, ριζοσπαστι... οι τάσεις ριζοσπαστικοποίησης και τα αίτια και οι ρίζες της ριζοσπαστικοποίησης να εντοπίζονται, να ταυτοποιούν κινούνται νωρί, έγκαιρα, ώστε να καταπολεμούνται έγκαιρα. Περί τίνο πρόκειται. Δεν πρόκειται για στιγματοποίηση ή δαιμονοποίηση. Πρόκειται πολύ περισσότερο για στοιχεία τα οποία θα πρέπει να μπορούν να εντοπίζονται το δυνατόν νωρίτερα, να ε, ε, ε το δυνατόν νωρίτερα ώστε προληπτικά να ερχόμαστε άμεσα σε επαφή με τα άτομα αυτά για να αντιμετωπίζουμε τις τάσεις ριζοσπαστικοποίησης ώστε ήδη εν τη γενέση να μπορούν αυτά, αυτές οι τάσεις να αντιμετωπίζονται, να αποφεύγονται. Νομίζω Πρόεδρε ε, μπόρεσα να καλύψω τα περισσότερα ερωτήματα. Αν δεν συμβαίνει αυτό πείτε το μου και στον επόμενο γύρο θα παρέμβω αντίστοιχα. Ευχαριστώ. Περνάμε σε επόμενη ομάδα ερωτήσεων. Παρακαλώ να είστε πολύ σύντομοι, λιγότερο από ένα λεπτό ο καθένας, για να προλάβουν όλοι. Ο κύριος Δίας Δημήρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ. Ειλικρινά, Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να εμπλέξουμε την ε, αστυνομία ε, εγκύτη την αστυνομία της γειτονιάς ε, σε θέματα ε, ριζοσπαστισμού ή σε θέματα σε προβλήματα τρομοκρατίας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το Κοινοβούλιο απέριψε πριν από μερικού μήνες το περίφημο πακέτο Europol. Ρωτώ λοιπόν... Αν πριν εξετάσουμε εν ώψη του 2013 την πρόταση κανονισμού αν αυτό το πακέτο Europol θα ξανάρθει εδώ στο Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε να το εξετάσουμε και με τους όρους της συνθήκης της Λισαβόνας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ γιατί είσαστε εδώ παρούσα σήμερα. Σημείωσα ότι αναφερθήκατε στο SIS-2, Schengen Information System 2 και σε σχέση και με τον προϋπολογισμό και το κόστος είχε γίνει συζήτηση και εδώ θα πρέπει να ενθαρρύνω εσάς να ενταχθεί το κόστος και ο προϋπολογισμός. Εδώ εμπλέκει το Κοινοβούλιο τους πολίτες και δεν κατανοούμε πώς ένα εγχείρημα το οποίο από το 2007 θα έπρεπε να λειτουργεί φτάνουμε στο 2010 και δεν υπάρχει κανείς που να καταφέρνει να καθορίσει ένα χρονοορίζοντα για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Και όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, είπατε ότι κατά τη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας κατά τον Οκτώβριο θα υπάρξει μια νέα πρωτοβουλία. Ελπίζω ότι θα είναι ένα χρονοδιάγραμμα ώστε το SIS, Schengen Information System, να είναι λειτουργικό το δυνατόν πιο νωρί. Αναφερθήκατε στην υπηρεσία μετά ή στην οργάνωση και ε, στον οργανισμό. Και έχω δύο ερωτήσεις εδώ. Όσον αφορά τον οργανισμό συμφωνούμε. Δεν είναι θέμα επίμαχο αυτό. Συμφωνούμε. Είναι ένας οργανισμός σημαντικός για να διαχειρίζεται τις τεχνολογίες της πληροφορίας σε αυτόν τον τομέα. Εντάξει, τώρα τι συμβαίνει όμως. Βλέπουμε ότι σε σχέση με τα, με τα κονδύλια περιέκοψε σημαντικά το Συμβούλιο την πρόταση που είχε υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να καταλάβω ποια είναι τα αίτια αυτή τη περικοπή από πλευρά του Συμβουλίου και αν η Βελγική Προεδρία εξακολουθεί να ακολουθεί αυτή την κατεύθυνση περικοπή, Τι θα γίνει σε σχέση με την υπηρεσία αυτή. Θα μειωθεί, θα συρρυκνωθεί το επίπεδο αρμοδιοτήτων τη. Μήπω θεωρείτε ότι μπορεί με λιγότερα χρήματα να λειτουργήσει εκείνο το οποίο πρέπει να κάνει η υπηρεσία αυτή. Και κάποια κράτη-μέλη φαίνεται ότι ενδιαφέρονται να αυξήσουν ε, με άλλες αρμοδιότητες αυτή την υπηρεσία, με νέες αρμοδιότητες. Ε, κατά τη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας θα υπάρξουν, κυρία Υπουργέ, προτάσεις να υπάρξουν νέα συστήματα που θα αυξήσουν τις αρμοδιότητες αυτής της υπηρεσίας ή θα παραμείνουμε με το ΣΥΣ, με το Eurodac και την και την διακόπτει ο και το ΒΙΣ ΣΥΣ uh, και Eurodac. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω από αυτά που είπε ο κύριος Καέγια με τον οποίο συμφωνώ απολύτως. Είμαι και σκιώδης εισηγήτρια για το συστήριο Ζήτησα από το συντονιστή της ομάδας μας ε, να κάνει μία ερώτηση όσον αφορά την υπηρεσία. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να μας δώσετε συγκεκριμένες πληροφορίες, όμως μας έχετε υποσχεθεί να ενημερώνετε το Κοινοβούλιο για τα όσα συμβαίνουν. Για άλλη μια πλευρά λοιπόν σας ζητώ να προσπαθήσετε να το κάνετε αυτό ειδικά τώρα που έχουμε αυτή την έκθεση, γιατί φοβάμαι ότι ορισμένοι λόγοι που ισχύουν για κάποιους από εμάς τους ευρωβουλευτές, ή τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, ότι αν ήταν ε, πιο σημαντικό το Στρασβούργο για τα όργανα ίσως θα έλυνε το δικό μας πρόβλημα να μην έχουμε δύο έδρες στο Κοινοβούλιο. Βεβαίως αυτό δεν είναι πρόβλημα τόσο του Συμβουλίου, ίσως της Επιτροπής. Εν πάση περιπτώσει παρακαλώ να μας κρατάτε ενήμερους. Ευχαριστώ η κυρία Μπορσαλίνο. όπως είπα και στον προκάτοχό σας ε, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε μια ιδιότυπη μορφή εγκλήματος τη μαφία η οποία κάθε φορά αλλάζει πρόσωπο και υπησέρχεται ολοένα και περισσότερο, παρισφρεί ολοένα και περισσότερο στην οικονομία με διάφορους τρόπους. Η Κομισιόν ε, με πληροφόρησε ότι υπάρχει μία οδηγία, θα υπάρξει μία οδηγία όχι μόνο για την κατάσχεση των ε, περιουσιακών στοιχείων ε, της μαφία αλλά και των της χρήσης αυτών των, ε, των χρημάτων που έχουν κατασχεθεί για κοινωνικά έργα. Θέλω επίσης να αναφερθώ και στους ε, μάρτυρες ε, στις δίκες κατά της μαφίας που είναι άτομα τα οποία διατρέχουν τεράστιους κινδύνους ξέροντας πολύ καλά ποιες είναι οι μέθοδοι. Λοιπόν, είναι προτεραιότητα ή δεν είναι προτεραιότητα όλα αυτά για την Βελγική Προεδρία. Ευχαριστώ. Τρεις ακόμη ερωτήσεις. Τέρεξ. Είχε πει ότι θέλει να ρωτήσει κάτι. Και μετά κύριος Μπρόνς. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρα. Συμφωνώ ότι είναι απαραίτητο να διακρίνουμε μεταξύ της διαφωνίας με αξίες με τις οποίες πάντα ανεχόμαστε και από την άλλη πλευρά την επιδίωξη αξιών όπως η βία ή η προτροπή βίας. Σήμερα χρησιμοποιείται ο ίδιος ε, αρνητικός όρος και για τις δύο μερικές φορές. Ορισμένες φορές αυτή η χρήση αμφίσιμων όρων είναι δείγμα του ότι δεν ξέρουμε ακριβώς που κινούμαστε και μπορεί να οδηγήσει δικαστικώς και σε αδικίες. Θυμηθείτε ότι όταν μιλάμε για την μη βία Έχουμε περιπτώσεις ε, λογοκρισίας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα την απαγόρευση κόμματος στο Βέλγιο και αντίστοιχη απειλή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι αλήθεια ότι η ελευθερία του λόγου δεν πρέπει να τηρείται όταν έχουμε προτροπή βίας, αλλά μόνο σε αυτή την περίπτωση. Οπουδήποτε αλλού υπερισχύει η ελευθερία του λόγου. Κυρία Αντζελίλη. Ε, ε, ευχαριστώ την Υπουργό. τη κάναμε ένα σωρό ερωτήσεις. Ε, εδώ, εδώ είμαι, λέει η κυρία Αντζελίλη και κουνάει το χέρι της. Λοιπόν, είπαμε πολλές ερωτήσεις, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε σε όλες. Θα ήθελα όμως να επανέλθουμε στην διακίνηση των ναρκωτικών και την αντιμετώπιση τους. Εγώ πιστεύω ότι πρόκειται για μια απόλυτη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ικανοποιήθηκα πλήρως από την απάντησή σας. Θα ήθελα επίσης να ξέρω ποια είναι η θέση της Βελγικής Προεδρίας ε, για, την, ε, για, τον, για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Και επίσης αυτό συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σε σχέση με το πρώτο θέμα που θα ξεκινήσω, το ΣΥΣ 2. Τι συμβαίνει. Στην συνάντηση του Οκτωβρίου από πλευρά Συμβουλίου υπήρξε συμφωνία σε σχέση με τον προϋπολογισμό και το περαιτέρω δρομολόγιο, διότι χρειαζόμαστε συγκεκριμένα αποτελέσματα και ήταν ε, διαρκή πολύ ε, το διάστημα και θα πρέπει να υπάρξει ένα δεύτερο ρώσιμο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Έχω την εντύπωση ότι όλοι οι μοχλοί χρησιμοποιούνται τώρα και δείχνουν προς την ορθή και ενιαία κατεύθυνση ώστε να έχουμε και τις σαφείς, τα σαφή πλαίσια για τον προϋπολογισμό. Όταν κάνουμε λόγο για αστυνομική συνεργασία και όταν κάνουμε λόγο για γενικά συνεργασία μέσα στο πλαίσιο της καταπολέμησης του διασυνοριακού εγκλήματος και εγκληματικότητας, χρειαζόμαστε ένα αντίστοιχο σύστημα πληροφόρησης και τραπεζών δεδομένων, διότι αυτή είναι η πεμπτουσία της συνεργασίας. Και μετά το Συμβούλιο της 5ης, 6ης ή 7ης Οκτωβρίου, δεν γνωρίζω ακριβώς πότε θα διεξαχθεί, οπωσδήποτε θα προσεγγίσουμε το Κοινοβούλιο για να αποσαφηνίσουμε ποιες προτάσεις θα βρίσκονται επί τραπέζης τότε όπως είπα, υπάρχει χρονοδιάγραμμα, θα υπάρξει χρονοδιάγραμμα, συγκεκριμένα δεδομένα για τον προϋπολογισμό και πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα. Το 2013 θα πρέπει να έχουν δρομολογηθεί τα μέτρα και να μπορούμε να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε, θα τα καταφέρουμε. Είναι προτεραιότητα για μας, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε με αξιόπιστο τρόπο να υπερασπιστούμε τις θέσεις μας. Ιδιαίτερα όταν θέλουμε λειτουργικοί να είμαστε, ε, όσον αφορά την καταπολέμηση του εγκλήματος και ε, δεν διασφαλίζουμε όμως ε, την πληροφορική συνιστόσα. Τώρα, για το δεύτερο θέμα δεν είναι καθόλου η καταστολή όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης. Δεν θέλουμε καθόλου να στιγματοποιήσουμε ή να δαιμονοποιήσουμε κάποιες στάσεις ή τοποθετήσεις. Αυτό που θέλουμε είναι και αξιωματικοί της αστυνομίας ασχολούνται ήδη με αυτό είναι με ορθό τρόπο να μπορέσουμε να ηχνηλατήσουμε, να ε, ταυτοποιήσουμε και εντοπίσουμε κάποιες ε, ε, τέτοιες τάσεις ώστε να αντιδράσουμε έγκαιρα και να δώσουμε έχουμε μια απάντηση έγκαιρα για τη ριζοσπαστικοποίηση. Είμαι πισμένη ότι οι αστυνομικές αρχές είναι εκείνες που πρέπει να μεριμνήσουν και να διασφαλίσουν ώστε σε μια σύντομη αρχική φάση να μπορέσουμε να δράσουμε. Δεν πρόκειται καθόλου για περιστολή της ελευθερίας της έκφρασης, αλλά πρόκειται για την καταπολέμηση των ριζοσπαστικών τάσεων από κοινού με συνεργασία με την κοινωνία, με street workers, με εργαζόμενους ε, που κατεβαίνουν για να συνεργαστούν με τους πολίτες ε, στους δρόμους και στις γειτονιές ε, και έτσι με συγκεκριμένο τρόπο μπορούμε να έχουμε ένα συγκεκριμένο εξειδικευμένο μέσο στα χέρια μας από πλευράς αστυνομίας για να δράσουμε σωστά. Είναι σημαντικό μέτρο για την αστυνομία ώστε η ριζοσπαστικοποίηση και οι τάσεις ριζοσπαστικοποίησης να μπορούν να καταπολεμηθούν έγκαιρα. Μετά, κοιτάζω βέβαια τώρα τις σημειώσεις μου για να μην ξεχάσω κάτι. Έτσι. Λοιπόν, ριζοσπαστικοποίηση, το κάλυψα το θέμα αυτό ήδη, μια στιγμή. Επόμενο, η Europol, η Ευρωπόλ ε, έγινε ερώτηση σχετικά. Δεν υπάρχουν άλλες συγκεκριμένες εξειδικευμένες πρωτοβουλίες που σχεδιάζονται υπό τη Βελγική Προεδρία. Θα παρακολουθήσω το θέμα βέβαια, αλλά και το Ευρωκοινοβούλιο θα διαδραματίσει το ρόλο του. Και ίσως σε μια ιστερότερη, μεταγενέστερη χρονική στιγμή θα ξανασυζητήσουμε το θέμα όταν θα έχουν προχωρήσει κάποια πράγματα. Τώρα για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Αυτό είναι προτεραιότητα ενωσιακά στην Ευρώπη για την ευρωπαϊκή κοινότητα. Υπάρχει και αυτό το σύμφωνο για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά πτυχών εδώ και συνιστοσών παραμέτρων που με άλλα λόγια θα μπορούσαν να ε, ληφθούν υπόψη και που πρέπει να εφαρμοστούν να εκτελεστούν συγκεκριμένες δράσεις και μέτρα. Πρέπει να εργαστούμε με αυτά που έχουμε στα χέρια μας και έχουμε μπροστά μας. Αλλά υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες. Αυτή η διασυνοριακή πτυχή που χαρακτηρίζει για παράδειγμα τα πυροβόλα όπλα, τα ε, ε, όπλα τα οποία χρησιμοποιούν ε, οι μετακινούμενοι κακοποιοί. Όταν ασχολείται κανείς με τα διασυνοριακά, με το οργανωμένο έγκλημα, φυσικά διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο το εμπόριο ναρκωτικών. Και σε σχέση με την προστασία μαρτύρων και προστασία ατόμων είναι αρμοδιότητα αυτό φυσικά των Υπουργών Δικαιοσύνης, των αρμόδιων για θέματα δικαιοσύνης. Είναι δύσκολο για μένα να τοποθετηθώ τώρα για αυτό το θέμα. Πρέπει όμως άνθρωποι οι οποίοι σε δίκες ε, έχουν να καταθέσουν ως μάρτυρες να προστατεύονται, να προστατεύονται αποτελεσματικά. Αλλά από την δικαιοσύνη πρέπει να καλυφθεί. Ε, Σας ευχαριστώ που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Είμαι σίγουρη ότι θα συνεχίσουμε τη συζήτηση και τη συνεργασία μετά τις θερινές διακοπές. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ερωτήσεις που απαντήσατε. Uh, Συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξη. Το επόμενο σημείο που βλέπω είναι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα PNR απολογισμός της αντιπροσωπείας της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ που πήγε στην Ουάσιγκτο. Θα ζητήσω από τη Σόφη που είναι η συγγήτρια, Σόφη Ιντεφέλτ, και η οποία ήταν και η επικεφαλής της αντιπροσωπείας να μας ενημερώσει σχετικά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να πω ότι θα σας παρέχουμε γραπτή έκθεση επί αυτής της σύντομης επίσκεψης, όμως να σας πω γρήγορα με ποιους συναντηθήκαμε, τι συζητήσαμε. Ήταν όντως πολύ σύντομη επίσκεψη, μόνο 48 ώρες. Το βασικό θέμα ήταν το National Targeting Center, το οποίο επισκεφτήκαμε και μας παρουσίασαν τις μεθόδους που χρησιμοποιούν κάναμε έναν σύντομο γύρο Επίσης συναντηθήκαμε με τον υπεύθυνο για την εσωτερική ασφάλεια, Homeland Security, με δύο μέλη του Κογκρέσου, διάφορους αξιωματούχους. Ορισμένοι από εμάς συναντήθηκαν και με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας επίσης με τον Αμερικανό πρέσβη κατά της τρομοκρατίας ενώ είχαμε και διάφορες συναντήσεις με think tank αλλά και με ακτιβιστές υπέρ της ε, ιδιωτικής ζωής και της προστασίας της. Δεν θα ήθελα τώρα να περάσω σε συμπεράσματα γιατί δεν έχουμε κάνει αξιολόγηση ως αντιπροσωπεία στην οποία αντιπροσωπεία συμμετείχα εγώ, οι σκιώδεις εισηγητές και ορισμένοι υπάλληλοι. Επαναλαμβάνω, δεν θέλω τώρα να μιλήσω για συμπεράσματα γιατί δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη ποια θα πρέπει να είναι αυτά τα συμπεράσματα νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τις πληροφορίες που λάβαμε σε σχέση και με το ψήφισμα που εγκρίναμε το Μάιο. Πρέπει λοιπόν να περιμένουμε και να δούμε το σχέδιο εντολής που ανακοίνωσε η Επιτροπή ότι θα δημοσιεύσει στις 7 Σεπτεμβρίου και το οποίο θα μας δώσει την διαπραγματευτική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έτσι περνάω στον δεύτερο μέρος ε, της ημερήσιας διάταξης για αυτό το σημείο η Ιαπωνία και ο Καναδάς μας έχουν ζητήσει να τους επισκεφθούμε, να κάνουμε μία αποστολή διακρύβωσης στοιχείων. Δεν ξέρω τι ισχύει από πλευράς ε, προϋπολογισμών, αλλά σας ενημερώνω. Και το δεύτερο κομμάτι του σημείου της ημερήσιας διάταξης αφορά την εφαρμογή εκ μέρους της Επιτροπής του ψηφίσματος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 2010. Όπως θα θυμάστε, στο ψήφισμα αναφερόταν προθεσμία για την συμμόρφωση όσον αφορά το πακέτο PNR μέχρι τον Ιούλιο, μέσα Ιουλίου δεν έχουν ε, κάνει κάτι εντός της προθεσμίας. Ε, τους γράψαμε λοιπόν για να τους ζητήσουμε να μας εξηγήσουν και θέλουμε να έρθουν εδώ στην Επιτροπή μας για να μην γίνει κάτι άτυπα. Άτυπα ακούσαμε ότι ένα μέρος του πακέτου για τα PNR θα το έχουμε στις 7 Σεπτεμβρίου. Αυτό όμως θέτει σε αμφισβήτηση το χρονοδιάγραμμα των συζητήσεων εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από τη μία πλευρά είναι αδικία να πιέζουμε χρονικά το Κοινοβούλιο, γιατί πάντα το Κοινοβούλιο μου φαίνεται καταλήγει να βιάζεται και να πρέπει να αποφασίσει εντός εβδομάδων μόνο, ενώ όλα τα άλλα όργανα πηγαίνουν με το πάσο τους. Καταλαβαίνω βεβαίως ότι ορισμένες φορές δεν υπάρχουν οι δυνατότητες από τα άλλα Λοιπόν, να επεξεργαστούν τα πάντα εντός λίγων εβδομάδων, αλλά και εμείς έχουμε τεράστιο έργο. Οπότε θα θέλαμε να ζητήσουμε από το Συμβούλιο να λειτουργήσει γρήγορα γιατί εμείς έχουμε δείξει ότι μπορούμε να σεβαστούμε σύντομες προθεσμίες και αν δεν γίνει κάτι τέτοιο μπορεί αυτό το πράγμα, το θέμα να λιμνάσει. Τέλος, θα ήθελα να ζητήσω δύο πράγματα από την Επιτροπή. Καταρχάς, μπορούμε να λάβουμε συγκεκριμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουμε θέσει επανειλημμένως στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο που έχουν αναφερθεί στα ψηφίσματα, που ήταν ερωτήσεις κοινοβουλευτικές και τα λοιπά. Θέλουμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Και τέλος, Μία ακόμη ερώτηση. Πριν ξεκινήσουν οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις, θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις για το τι ισχύει Ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά τις διμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ κρατών μελών και ΕΠΑ για την άρση υποχρέωσης θεώρησης. Θα θυμάστε όσοι ήσασταν και παλαιότερα στην Επιτροπή ότι σε αυτές τις διμερείς διαπραγματεύσεις στις οποίες δεν έχει καμία ανάμειξη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν γνωρίζουμε τι αφορούν αυτές τις διαπραγματεύσεις. Το μόνο που γνωρίζουμε ήταν ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είχαν μια σειρά από προϋθέσεις που θα έπρεπε να τηρούν τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη και μία προϋπόθεση ήταν η υποχρέωση για δεδομένα PNR, δεδομένα των επιβατών. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα μπορέσουμε να ρυθμίσουμε αυτό το θέμα ταυτόχρονα και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Σόφη. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη γραπτή έκθεση και την αξιολόγησή σας. Όπως είπε και η Σόφη, στο ψήφισμα της 5ης Μαΐου ζητήσαμε από την Επιτροπή να παρουσιάσει την πρόταση της το αργότερο μέσα Ιουλίου. Όμως από ό,τι γνωρίζουμε δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής, οπότε θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Αλμέιντα να μας πει πώς εξελίξονται τα πράγματα. Καλό σας απόγευμα, αγαπητά μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ Πολιτικών Ελευθεριών. Είμαστε απασχολημένοι και ασχολούμαστε με την εκπόνηση των διαδικασιών για το πρώτο πακέτο PNR σε σχέση με το Σεπτέμβριο. Έχουμε ολοκληρώσει τις εσωτερικές διαβουλεύσεις ε, διυπηρεσιακά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να έρθουμε σε επαφή και με άλλες υπηρεσίες πέρα από την Διεύθυνση Εσωτερικών ε, Υποθέσεων σε σχέση με τις απόψεις ε, για το PNA. και επαναλαμβάνω στις 7 Σεπτεμβρίου αναμένουμε να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε σε εσά και στο Συμβούλιο τρεις διαπραγματευτικές εντολές με τις ΗΠΑ, με την Αυστραλία και τον Καναδά και μια ανακοίνωση, μια ευρύτερη γενικότερη ε, ανακοίνωση για το πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε το PNR να διαφοροποιείται ή να προσαρμόζεται ώστε να έχουμε μια ενιαία πολιτική σε σχέση με ε, κυρίαρχα κράτη που θα θέλουν να έρθουν σε διαπραγματεύσεις μαζί μας και να ακολουθηθεί μια ενιαία κατεύθυνση. Ξέρουμε ότι η Νότια Κορέα πριν από την ε, υιοθέτηση της συνθήκης Λισαβόνας ήθελε να υπάρξει μια συμφωνία και αρνηθήκαμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις λόγω των θεσμικών μεταβολών που θα ίσχυαν και η Ιαπωνία ήταν σε στενή επαφή μαζί μας για τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις. Θεώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρειάζεται μια γενικότερη, σφαιρικότερη πολιτική και κατευθύνσεις ε, επί των οποίων θα είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε θέματα με τρίτες ε, χώρες και όχι να ακολουθήσουμε μια τυχαία συγκυριακή πολιτική για το πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αιτήματα τέτοιων χωρών. Στο Σεπτέμβριο, 7 Σεπτεμβρίου θα έχετε αυτή τη γενική ε, ανακοίνωση για αυτή την ε, εντολή και για την διαφοροποιημένη τοποθέτηση σε σχέση με τον ε, Καναδά, την Αυστραλία και τη ΣΥΠΑ. Υπάρχει μια χασμοδία έναντι του Καναδά και αν δεν καλυπτόταν αυτό το χάσμα, αυτό το κενό θα είχαμε προβλήματα λόγω για παράδειγμα της ε, συνθήκης ε, της ε, νίκαιας για παράδειγμα σε σχέση με εξουσίες και αρμοδιότητες που δεν έχει το Κοινοβούλιο όπως υπό τη συνθήκη της Λισαβόνας για παράδειγμα για την σφαιρική συμφωνία που θα ρυθμίζει τέτοιου είδους μεταφορές δεδομένων όσον αφορά τον Καναδά. Τέτοιου είδους ε, δεσμεύσεις από πλευράς ε, του Καναδά θα πρέπει να θεωρηθούν ε, επαρκείς για την διαβίβαση από και προς τον Καναδά. Με την Αυστραλία και τις ΗΠΑ έχουμε προσωρινά ισχυρές τέτοιες συμφωνίες που έχουμε διαπραγματευτεί υπό την συνθήκη της Νίκαιας. Τώρα όμως, μια και δεν ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του Ευρωκοινοβουλίου όσον αφορά τις διευρυμένες αρμοδιότητες της συνθήκης Λισαβόνας έχει προσαρμοστεί, έχει αλλάξει η εντολή ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η ε, διαπραγμάτευση αυτών των ε, εντολών με πλήρη υποστήριξη κοινοβουλευτική. Για το δεύτερο τμήμα τώρα του ε, πακέτου που καθυστέρησε μέχρι την έναρξη του 2011 διότι οι εσωτερικές διαπραγματεύσεις μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέδειξαν ότι χρειαζόταν μια νέα μελέτη επιπτώσεων ώστε να ε, τεκμηριωθούν και να ε, ε, υποστηριχθούν οι προτάσεις PNR και Χρειαζόμαστε μια τέτοια εξέταση και ανάλυση των ε, μελετών επιπτώσεων μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε σχέση με αυτά τα οποία αρχικά ε, είχαμε σχεδιάσει για τις ε, εντολές αυτές σε σχέση με την πρόταση για το PNA δεν θα υπάρξει η τριχοτόμηση αυτή αλλά θα σας δώσουμε την ανακοίνωση το Σεπτέμβριο και ελπίζουμε την πρόταση PNR κατά την αρχή του 2011 ενωρίς σχετικά. Γνωρίζω ότι η κυρία Εντεφέλτ έχει ζητήσει επανειλημμένα σε σχέση με την ερμηνεία που έχει δοθεί όσον αφορά αμερικανικό νομοθέτημα το οποίο ε, εγκρίθηκε σε σχέση με τα θέματα PNR τον Φεβρουάριο και μια ε, τροποποίηση προσαρμογή του Privacy Act όσον αφορά την διαβίβαση αυτών των στοιχείων έχω την εντύπωση ότι η Επίτροπος Μάλμστρομ με βάση πληροφορίες που είχαν δοθεί σε εκείνη στο γραφείο της για την άποψη την περιερμηνίας άποψη από πλευράς μας από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίπτωση αυτή κατά τα άλλα θεωρούμε ότι οι οι οποίες έχουν διαμορφωθεί λαμβάνουν υπόψη όλα τα θέματα τα οποία εσείς ζητήσατε στο ψήφισμά σας να διασφαλιστούν. Ελπίζω λοιπόν ότι η νέα πολιτική μας ε, για τα PNA θα ξεκινήσει με πλήρη κοινοβουλευτική υποστήριξη από το Σεπτέμβριο και εφ' Ευχαριστώ, ελπίζω να μην χρονοβόρησα. Thank you very ε, Ευχαριστώ. Άρα 7 Σεπτεμβρίου μπορούμε να αναμένουμε μια γενική ανακοίνωση. Ένα άλλο ερώτημα τέθη όσον αφορά τις ε, διμερείς αυτές συμφωνίες ε, άρσης υποχρέωσης θεωρήσεων και τον συσχετισμό της ε, με τα δεδομένα PNR. Μπορείτε να απαντήσετε τώρα δεν είμαι υπεύθυνο για αυτό το κομμάτι της πολιτικής μας, την άρση υποχρέωσης θεωρήσεων. Θα πρέπει να συζητήσω με τους συναδέλφους για να απαντήσω πλήρως στην κυρία Ιντεφέλτ. Θα διαβιβάσω όμως την ερώτηση. Δύο ερωτήσεις. Φως, παρακαλώ. Δεν ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να πω το ίδιο το πρόγραμμα στη ΣΥΠΑ ήταν έντονο, ήταν καλό και θα ήθελα να ευχαριστήσω ταυτόχρονα για την καλή ηγεσία της κυρίας Ιντφέλτ. Καλά τα πήγε τα πράγματα σε σχέση με την ε, επικεφαλή επικεφαλής της αντιπροσωπείας. Χωρίς να θέλω να προδικάσω για την αξιολόγηση στην ομάδα μας και στην ομάδα σκιωδών εισηγητών σίγουρα θα ξανασυζητήσουμε αυτά τα θέματα όμως τα συμπεράσματα που κατάφερα να αποκομίσω είναι ότι ουσιαστικά το PNR είναι κάτι το καλό για τις πληροφορίες που μπορούν να διαβιβαστούν και είναι κάτι το θετικό λοιπόν που αξίζει να αντιμετωπιστεί σε βάθος. Με ενδιαφέρον θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της διάρκειας της αποθήκευσης στοιχείων και θα ξανασυζητήσουμε το θέμα με, το, με τη μέθοδο push ή pull δηλαδή ε, για το πώς θα αντλούνται αυτά τα στοιχεία μετά από αίτημα και για τον εκπρόσωπο εκπρόσωπο της Επιτροπής σε σχέση με το θέμα της χρονικής διάρκειας, βλέποντας το SWIFT και το PNR, φυσικά ε, ε, διαφέρουν όσον αφορά την γενική προσέγγιση. Εκείνο το οποίο είναι ουσιώδες όμως είναι η διαβίβαση στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη ΣΥΠΑ. Η διαβίβαση στοιχείων από την Ευρώπη στη ΣΥΠΑ. Και οι προδιαγραφές προστασίας ε, δεδομένων θα πρέπει να προσεχτούν. Για το το SWIFT μπορούμε να καταλήξουμε, καταλήξαμε γοργά σε ένα αποτέλεσμα. Όμως ελήψη κοινών προδιαγραφών για το PNA κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να υπάρξει κάποια καθυστέρηση και ίσως δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πιο γοργά γιατί για τη διαβίβαση στοιχείων ένας ε, παρόμοιος τομέας ε, ή και μια ας το πω έτσι ανάλογη κατάσταση διαμορφώνεται όπως το SWIFT. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Είναι σημαντικό να δούμε αυτό το συσχετισμό μεταξύ αυτών επίσης. Και άλλα σχόλια ή ερωτήσεις από τον κύριο Κέρκοπ και η κυρία Λάτφορντ. Ευχαριστώ. και από πλευρά ε, των σχεδόν εισηγητών. Θα ήθελα να ε, συγχαρώ και εγώ την Σοφίντ για τον ηγετικό της ρόλο σε αυτή την αποστολή στις ε, ΗΠΑ και σε σχέση με τη σημερινή τοποθέτηση για το πώς καταλήγουμε σε αυτά τα αποτελέσματα θα ήθελα απλά και μόνο να πω το εξής, να αναφερθώ στην Συμφωνία PNR, διότι όπως γνωρίζουμε Υπάρχουν αρκετές ε, συμφωνίες PNR με διαφορετικά νομοθετικά πλαίσια έναντι διαφορετικών χωρών και έναντι των διαφορετικών θεμάτων που αντιμετωπίζουμε για τη χρήση δεδομένων, για την προστασία των ατόμων και των, ε, της ιδιωτικής, ιδιωτικής τους ζωής και την διάρκεια καταχώρησης πληροφοριών είναι εκπληκτικό ότι οι προδιαγραφές είναι τελείως διαφορετικές όσον αφορά όλα αυτά τα πλαίσια. Έχουμε μια κατάσταση όπου όλοι θεωρούν ότι η δική τους αντιμετώπιση για τα δεδομένα είναι η πιο ασφαλής ε, και η πιο ε, σίγουρη. Έχουν επιχειρήματα ίσως για κάποια τέτοια τοποθέτηση, αλλά έχουμε και εμείς τις δικές μας προδιαγραφές. Και το θέμα είναι ότι εξετάζοντας τις διάφορες συμφωνίες μπορούμε να βρούμε κοινού παρονομαστές, κοινά στοιχεία που θα μας επιτρέψουν επιτρέψουν να καταλήξουμε σε συμφωνίες χωρίς κάθε συμφωνία να είναι τόσο ξεχωριστή και μοναδική που να είναι πολύ δύσκολο να διασφαλιστεί μέσα σε μια κοινή βάση η προστασία αυτών των δεδομένων. Πολύ προσπάθεια πρέπει να γίνει για να καταλήξουμε σε έναν ε, κοινό παρονομαστή και μια προσέγγιση κοινών στοιχείων ώστε οι προδιαγραφές που θα εφαρμόζονται θα είναι οι ίδιες κοινέ προδιαγραφές παρότι θα παρέχονται αυτά τα στοιχεία σε διαφορετικές χώρες με διαφορετικά νομοθετικά πλαίσια διαδικασία και διαφορετικές, διαφορετικά συντάγματα και συνταγματικές διατάξεις. Αυτό είναι κάτι το πολύ ενδιαφέρον, όχι μόνο όσον αφορά το PNR, αλλά και τις συμφωνίες πλαισίου που θα αντιμετωπίσουμε πολύ σύντομα. Αυτό το οποίο αποκομίσαμε από την επίσκεψη στη ΣΥΠΑ, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι ΙΠΑ πιστεύουν ότι έχουν υψηλότατες προδιαγραφές. Ε, το ότι δεν ε, προσαρμόζονται απόλυτα και δεν έχουν απόλυτα συμβατές ε, διατάξεις όσον αφορά εκείνες της Ευρώπης είναι κάτι προφανές και αυτό οδηγεί σε ελέγχους στα σύνορα κτλ. Λοιπόν, αυτό θα το δούμε πάρα πολύ προσεκτικά και υποστηρίζω πάρα πολύ αυτό το οποίο αναφέρθηκε από τον κύριο Φως Υπάρχει θέμα πρόσθετης αξίας εδώ, σίγουρα από την παροχή πληροφοριών και την καλή και υπεύθυνη χρήση αυτών των πληροφοριών. Είναι σημαντικό στοιχείο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διεθνούς τρομοκρατίας. Και εμείς όμως έχουμε δουλειά ως κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των πολιτών μας να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της προσέγγισης των αρχών και των δικαιωμάτων των πολιτών. Και πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την προσέγγιση να διασφαλιστεί αυτή η ισορροπία καθώς συνεχίζουμε το έργο μας. Ευχαριστώ. Από ό,τι βλέπω από αυτή την επίσκεψη προέκυψαν ακόμη περισσότερα ερωτήματα όσον αφορά τον κοινό παρανομαστή για την προστασία δεδομένων. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε απαντήσεις λοιπόν επί των βασικών ενιών. Κυρία Λάτφορντ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρα. Η απάντηση της Επιτροπής με άφησε λίγο ενοχλημένη για δύο λόγους. Καταρχάς, είπατε ότι δεν είστε αρμόδιοι για τις ε, άσεις υποχρέωσης θεωρήσεων στα PN και τα PNR δεν μου φαίνεται καλή απάντηση γιατί ρωτήσαμε τι γίνεται όσον αφορά τις διμερείς διευθετήσεις για τα PNR στα πλαίσια των διμερών συμφωνιών για τις θεωρήσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι σχετικό θέμα και σχετίζεται και με την ανακοίνωση που αναβλήθηκε για το Σεπτέμβριο. Κάποια στιγμή λοιπόν, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, πρέπει να λάβουμε κάποιες διευκρινήσεις από αυτού. Και το δεύτερο σημείο, ε, το έχω ξεχάσει, ελπίζω ότι θα μας ενημερώσει η Σόφη, ποια είναι η νομοθετική αλλαγή στις Ηνωμένε Πολιτείες. Όμως, όταν ε, το θέτει το θέμα δημοσίως η συγγήτρια στην Επιτροπή, ευελπιστεί και σε μια δημόσια απάντηση. Δεν ξέρω αν η Σόφη έχει λάβει απάντηση από την Επιτροπή και μπορεί να μας ενημερώσει σχετικά. Όμως δεν μας ικανοποιεί καθόλου το γεγονός ότι δεν λαμβάνουμε απαντήσεις και μας λέτε θα σας απαντήσουμε αργότερα. Ευχαριστώ κύριο Σταβάρες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι σχετικά καινούριο και δεν ήμουν ο αρχικός σκιώδης εισηγητής της ομάδας μου, άρα θα περιοριστώ στο να πω ότι ήταν ενδιαφέρουσα η επίσκεψη στην Ουάσιγκτον. Για παράδειγμα είδαμε πού γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων PNR, μια δυνατότητα που δεν είχαμε στην περίπτωση του SWIFT Δηλαδή οι Ηνωμένε Πολιτείε μας ζητάν τα δικά μας δεδομένα, αλλά δεν μας εμπιστεύονται ούτε καν για να μας δείξουν τις εγκαταστάσεις τους. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω την Σόφη για το έργο της και για τον ειλικρινή και πολύ επικοδομητικό τρόπο με τον οποίο συνεργάστηκε με τους συζητητές. και βεβαίως ε, αναμένουμε με ανυπομονησία την εντολή. Σόφη, θες να απαντήσεις. Ναι, πολύ σύντομα να συνοψίσω. Να πω και πάλι στην Επιτροπή ότι εμείς ως Κοινοβούλιο ομοφόνος προσπαθούμε να σας βοηθήσουμε και να προχωρήσουμε. Και με απογοητεύει λίγο ότι πρέπει να τραβάμε με το ζόρι κάθε κομματάκι πληροφορίας από την Επιτροπή και το Συμβούλιο και νομίζω ότι δεν έχω λάβει επίσημη απάντηση στην ερώτηση που είχα κάνει. Έχω λάβει άτυπη απάντηση, έχω λάβει και άτυπες απαντήσεις από διάφορες νομικές υπηρεσίες, αλλά διαφέρουν μεταξύ τους και θέλω μια επίσημη νομική απάντηση μάθαμε στην Ουάσιγκτον ότι είχαν προταθεί αλλαγές τον Αύγουστο του 2007, ένα μήνα μετά την συμφωνία. Αυτοί μας είπαν ότι ήταν φυσιολογικές αυτές οι αλλαγές μετά την έγκριση μιας συμφωνίας, ενώ οι δικές μας ε, νομικές υπηρεσίες μου λένε ότι δεν είναι συμμόρφιο με την συμφωνία αυτή διαδικασία. Θέλω μία απάντηση. Έχουμε βάλει τις ερωτήσεις μας και στα ψηφίσματα. Κάποιος ας μας εξηγήσει. Γιατί δεν επαρκούν τα δεδομένα PNR εδώ. Θέλουμε μία κανονική απάντηση, όχι να μας το εξηγείτε κάπου. Ζητάμε απαντήσεις από το 2003. Δεν είναι καινούργια αυτά τα θέματα το θέμα της, ε, των συμφωνιών ε, άρσης υποχρέωσης θεωρήσεων. Και τα έχουμε βάλει τόσες φορές στα ψηφίσματα. Κοιτάξτε, προσπαθώ να γίνω καλή και δεν μου βγαίνει και από φυσικού μου. Θυμάστε τι είχε γίνει και με τις διαπραγματεύσεις για τις θεωρήσεις. Πριν από δύο χρόνια είχαμε αποφασίσει να έχουμε μία παράλληλη προσέγγιση. Από τη μία πλευρά διαπραγματεύσεις της Επιτροπής, από την άλλη διαπραγματεύσεις των κρατών μελών. Γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείες δεν δέχονται ότι η Ευρώπη μιλάει με μία φωνή. Αυτό είναι κακό από μόνο του. Και είχαν και αυτή τη λίστα με τις προϋποθέσεις προκειμένου τα κράτη-μέλη να κρατήσουν ή να αποκτήσουν την άρση υποχρέωσης θεωρήσεων που συμπεριλαμβάνει αυτή η λίστα επιπλέον μέτρα ασφαλείας στα αεροδρόμια αλλά και πρόσβαση στα αστυνομικά δεδομένα, σε δεδομένα DNA, σε δεδομένα πινακίδων κυκλοφορίας, σε δεδομένα απορριφθέν των αιτήσεων προσφυγών και δεν ξέρω, ενδεχομένω να θέλουν και πρόσβαση στο Eurodac και τα λοιπά. Και βεβαίως σας υπενθυμίζω ότι έχουν και πρόσβαση στα δεδομένα μας που έχουν εταιρείε που βασίζονται, που έχουν έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι άλλο παραπάνω θέλουν δηλαδή θέλουμε κάποιες απαντήσεις σε απλά ερωτήματα. Είναι υπερβολικά αυτό. Σας βάλαμε μια προθεσμία μέσα Ιουλίου. Δεν καταφέρατε να την τηρήσετε. Μπορείτε να μας απαντήσετε σε αυτά τα ερωτήματα που έχουμε θέσει τόσες φορές. Μπορούμε να λάβουμε μια υπόσχεση από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή ότι αν έχουμε την ανακοίνωση 7 Σεπτεμβρίου θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία πριν το τέλος του έτους. Αυτά και θα ξαναγίνω καλή τώρα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι τι ίδιε εμπειρίες έχουμε και με την συμφωνία SWIFT. Όταν μίλησε με μία φωνή η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν πολύ πιο ανοιχτές οι Ηνωμένε Πολιτείε όσον αφορά τις προϋποθέσεις και νομίζω ότι το ίδιο μοντέλο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και για τα δεδομένα PNR. Κύριε Αλμέιντα παρακαλώ. Θα προσπαθήσω να γίνω συμπαθητικός, όσο πιο συμπαθητικός μπορώ. Για το ερώτημα του κυρίου Φως για το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές διατάξεις προστασίας δεδομένων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όντως ισχύει αυτό και γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Θα μου πείτε γιατί να μην κάνουμε μία φορά μόνο διαπραγματεύσεις και να καταλήξουμε σε μία γενική συμφωνία επί της προστασίας δεδομένων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έτσι να ολοκληρώσουμε με αυτό το θέμα και να μην έχουμε τις ίδιες διαπραγματεύσεις κάθε φορά που μιλάμε για νέο σύστημα ανταλλαγής ε, προσωπικών δεδομένων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι και τα δύο χρειάζονται. Και ένα γενικό πλαίσιο που να δίνει τις βασικές αρχές με τις οποίες ε, Ευχαριστώ συμμορφώνονται και οι δύο πλευρές του Ατλαντικού, αλλά υπάρχουν και κάποια θέματα που πρέπει να αφορούν συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις. Για παράδειγμα, όταν στέλνουμε δεδομένα για ένα συγκεκριμένο σκοπό, δεν μπορούμε να μιλάμε έτσι αφηρημένα για το πόσο θα πρέπει να διατηρηθούν αυτά τα δεδομένα, χωρίς να γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο σκοπός χρήσης τους. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν θα μπορούσε ποτέ να επιληθεί. Θα μας έλεγαν ότι ένα γενικό πλαίσιο δεν θα μας έλεγε πόσο πρέπει να κρατηθούν τα δεδομένα από τις διάφορες υπηρεσίες ή από την αστυνομία. Γιατί κάθε φορά πρέπει να διατηρούνται για όσο είναι απαραίτητο και το πόσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο είναι κάτι το οποίο αποφασίζεται κάθε φορά σε συγκεκριμένες ξεχωριστές διαπραγματεύσεις. Και τώρα θα ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις για τα PNR βεβαίως από το Σεπτέμβριο. Τώρα, ε, περνάω στον κύριο Κέρκχοπ. Ναι, όντω χρειαζόμαστε έναν κοινό παρανομαστή. Θέλουμε να έχουμε μια γενική πολιτική που θα μας δίνει τις γενικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι διατεθειμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαπραγματευτεί με άλλα κράτη ή οντότητες. Χωρίς πολλές εξειδικευμένες διατάξεις. Ένα μοναδικό πλαίσιο βασικών αρχών με το οποίο θα συμμορφωνόμαστε. Γιατί να τώρα έχουμε Ηνωμένε Πολιτείε και Καναδά ως εταίρους με τους οποίους έχουμε διαπραγματεύσεις, αλλά δεν ξέρουμε ποιες ακόμη χώρες θα μας ζητήσουν δεδομένα PNR τα επόμενα 5-6 χρόνια. Και μπορεί να προκύψουν και εκπλήξεις. Όσον αφορά τώρα τις διμερείς διευθυντήσεις για την άρση υποχρέωσης θεωρήσεων. Με συγχωρείτε που γίνομαι ενοχλητικός, αλλά δεν μπορώ να σας δώσω την κατάλληλη απάντηση. Θα διαβιβάσω τις ανησυχίες σας στην Επιτροπή και σύντομα θα λάβετε μια σωστή απάντηση. Εγώ όμως δεν έχω όλες τις πληροφορίες, δεν έχω όλη την εικόνα μπροστά μου, όπως θα περιμένατε να λάβετε από εμένα όσον αφορά τις αλλαγές ε, στην νομοθεσία για την ιδιωτική ζωή φέτος. Με ενημερώνουν οι υπηρεσίες μου ότι ο στόχος αυτής της νομοθετικής μεταρρύθμισης της Αμερικανικής είναι να υπάρξουν εξαιρέσεις στο νόμο για δικαιώματα που έχουν οι πολίτες που είναι αρκετά παρόμοια αν όχι ταυτόσιμα με τις περιορισμούς που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ε, λόγους, αιτίες ε, τήρησης δημόσιας τάξης. Έτσι η αστυνομία δεν είναι υποχρεωμένη να δίνει δεδομένα και πληροφορίες για τους ε, εγκληματίες για τους οποίους έχει στοιχεία. Και αυτό είναι ταυτόσιμο και στις Ηνωμένε Πολιτείες υπάρχουν αυτές οι εξαιρέσεις που ισχύουν στο σύστημα δημόσιας τάξης. Θα ζητήσω πάντως από την Επιτροπή να σας σταλούν αυτές οι πληροφορίες επισήμως και όχι ανεπισήμως όπως από ό,τι φαίνεται έχει γίνει. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, πάλι θα διαβιβάσω τα μηνύματα ενόχλησης που άκουσα σήμερα και που έχω ακούσει αρκετές φορές αλλά για τα οποία δεν μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή κάτι. Ευχαριστούμε για τις απαντήσεις και ελπίζουμε να λάβουμε απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα στο εγγύς μέλλον. Ευχαριστούμε λοιπόν και συνεχίζουμε με την ημερησία διάταξη. Περνάμε στην ενημέρωση σχετικά με τις διαξαγόμενες διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες επανιστοχής. Αυτή η συζήτηση θα γίνει και κλεισμένων των θυρών. Όποιος λοιπόν ανήκει στο κοινό παρακαλώ να βγουν από την αίθουσα.